Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω θερμά. Είχα μία συνάντηση με τον Τούρκο πρέσβη οποίος με ενημέρισε ε, για την ε, κατάσταση στην ε, Συρία και όχι για την Κύπρο και λέω όχι δεν μιλήσαμε για την Κύπρο γιατί με τσιγκλάει ο κύριος Κασουλίδης και ε, σχετικά με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σχετικά με τα σύνορα της ε, Συρίας βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια αλληλεγγύη και σχετικά με τον αριθμό των προσφύγων οι Ευρωπαίοι έχουν ευαισθητοποιηθεί και πρέπει να παρακολουθούν τι γίνεται στα ε, κράτη-μέλη και να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε διότι ότι ε, χθε αποφασίσαμε στο διευρυμένο Προεδρείο ότι του χρόνου μία αντιπροσωπεία της ΑΦΕΤ θα πάει στην Τουρκία. Ακριβώς ε, ε, νομίζω λοιπόν ότι αυτό το πρόβλημα ήταν ένα κατάλληλο μήνυμα στην κατάλληλη στιγμή και θέλω να τονίσω εδώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για, από πλευράς τουρκικής και ευρωπαϊκής ε, ε, για τους ε, για την παρούσα κατάσταση. Ε, θεωρώ ότι η Τουρκία είναι πολύ σημαντική γεωγραφικά αυτή τη στιγμή και όλα τα θέματα πρέπει να τα χειριζόμαστε πάρα πολύ προσεκτικά. Χαίρομαι ότι θα καλύψουμε με τον Γενικό Γραμματέα της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών ε, Σχέσεων το θέμα αυτό και χαίρομαι χαίρομαι ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για την Συρία, για την κατάσταση στα σύνορα της Συρίας προς Λίβανο, προς Ιορδανία, ε, τις σχέσεις ε, ε, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε για να καταλήξουμε σε μία θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και για τα θέματα που άπτονται του αεροπλάνου με πολεμικό υλικό το οποίο ε, εχθές ε, κρατήθηκε από την Τουρκία και όπου πιστεύω ότι η κίνηση αυτή ήταν πολύ σωστή ε, εξού και θα χαρώ ιδιαιτέρως εάν ο κύριος Βημό μπορεί να μας πει εδώ τι γίνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο στα προκαταρκτικά μου σχόλια, διότι νομίζω ότι αυτό που έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι να μου θέσουν ερωτήσει ε, τα μέλη του Κοινοβουλίου και να κάνω και μια απόπειρα να απαντήσω φυσικά αν μπορώ. Να σα ενημερώσω λίγο λοιπόν για την κατάσταση, λαμβάνοντα υπόψη ότι η ύπατη εκπρόσωπος είχε έρθει την Τρίτη, επομένως ε, έχετε λάβει μια πλήρη εικόνα και περιγραφή του τι ακριβώς συμβαίνει, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε μια διαφορετική διάσταση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Και κυρίως να σας ενημερώσω, διότι δεν θα ήθελα να αναφέρω όλα τα στοιχεία τα οποία γνωρίζετε ήδη πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πιο πιεστικό ζήτημα στο όλο θέμα είναι η ανθρωπιστική κατάσταση, και η ανθρωπιστική βοήθεια. Όπως γνωρίζετε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε δεσμεύσει επιπλέον 50 εκατομμύρια προκειμένου να συνδράμουμε τους πρόσφυγες και τον εκτοπισμένο πληθυσμό στη Συρία οι οποίοι πλέον αριθμούν πάνω από 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, τεραστίων διαστάσεων για όλους μας. Και προ το παρόν υπάρχουν διάφορες ιδέες τις οποίες ίσως γνωρίζετε, αλλά μία που κυριαρχεί είναι μία ιδέα που εμφανίζεται μεταξύ κρατών μελών ε, για να δούμε πώς μπορεί να σταλεί απευθεία ε, η βοήθεια στου ανθρώπου εντό τη χώρα. Το μεγαλύτερο τμήμα τη ανθρωπιστική βοήθεια προσφέρεται στου πρόσφυγε στα σύνορα. Και ο, ο πρόεδρο σα ανέφερε προηγουμένω το Λίβανο, την Ιορδανία, ακόμα και το Ιράκ και την Τουρκία. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε ε, να συνδράμουμε και τον πληθυσμό ο οποίος βρίσκεται εντός της Συρίας, όπου βεβαίως η κατάσταση είναι τέτοια ώστε να περιπλέκει τη δυνατότητά μας να φτάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Εξετάζουμε λοιπόν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις τοπικές αρχές ή τις τοπικές κυβερνήσεις σε κάποιες από τις απελευθερωμένες περιοχές, να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε πιο ασφαλή νοσοκομεία και να μπορούν να εργάζονται με καλύτερο τρόπο. Κάποιες ε, κυβερνήσεις έχουν παρουσιάσει κάποιες ιδέες, υπάρχουν και συζητήσεις εν εξελίξει στον ΟΗΕ και βεβαίως το θέμα θα αναφερθεί και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ε, τη Δευτέρα από κάποια κράτη-μέλη. Εμείς, ε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με τους φίλους μας από την ΕΚΟ και από την ΕΦΚΟ εξετάζουμε το θέμα πολύ προσεκτικά και το εξετάζουμε και από νομική σκοπιά, ε, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τα διάφορα χρηματοοικονομικά ζητήματα, τον κανονισμό ή οποιονδήποτε άλλο περιορισμό υπάρχει στο συγκεκριμένο τομέα. Όσον αφορά τώρα το πώς έχει η παρούσα στρατιωτική κατάσταση ε, και ποιες ε, περιοχές τελούν υποκατοχή, Υπάρχει αυτή η διάσταση μεταξύ Συρίας και Τουρκίας, η οποία συνεχίζεται εδώ και μια εβδομάδα. Δεν έχει συμβεί τίποτα συγκεκριμένο την τελευταία ημέρα, αλλά οι τουρκικές αρχές εξηγούν με ιδιαίτερο σένος ότι δεν θα επιτρέπουν ε, πλέον στον ε, Συριακό στρατό να ε, εισβάλλει στην τουρκική επικράτεια. Οι τουρκικές αρχές ε, έχουν λάβει και ε, στήριξη από τον ΝΑΤΟ, από τα Ηνωμένα Έθνη και φυσικά ε, προσέχουμε την εξετάζουμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά. Όσον αφορά το θέμα των κυρώσεων, για το τι συνέβη εχθές σε ένα τουρκικό αεροδρόμιο, ένα αεροσκάφος σταμάτησε, προσγειώθηκε σε ένα τουρκικό αεροδρόμιο και επιθεωρήθηκε για όπλα. Και μία ε, πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης είναι ότι οι εθνικές αρχές μπορούν όταν επιβάλλονται κυρώσεις να εξετάζουν πώς εφαρμόζονται ε, τα διάφορα θέματα, αλλά πρέπει να δούμε από εκεί και πέρα και τι ισχύει και στην ε, τουρκική νομοθεσία και τι μπορεί να γίνει από αυτή την πλευρά. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που είδαμε και εμείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, για τον εξοπλισμό, ο οποίος κατασχέθηκε από το αεροσκάφος. Ε, ίσως τις επόμενες μέρες θα μάθουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, ένα τελευταίο για τις κυρώσει Θα υπάρχει ένα επιπλέον ε, ε, πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τη Δευτέρα, αλλά ακόμα υπάρχει προετοιμασία και αύριο ή σήμερα θα συζητηθεί και στην Κορεπέρ συμπεριλαμβάνονται ε, κάποια στοιχεία για απαγορεύσεις θεωρήσεων, ε, ε, πάγωμα στοιχείων ενεργητικού και θα δούμε αν υπάρχει δυνατότητα για άλλες κυρώσεις, θα δούμε αν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον κυρώσεις, διότι ούτως ή άλλως υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ε, κυρώσεων, ο οποίος έχει αρχίσει να επιβάλλεται από πέρσι. Όσον αφορά τώρα την αντιπολίτευση, ε, να σας πω ότι υπάρχει μία πρωτοβουλία την οποία παρακολουθούμε πολύ στενά, που είναι η πρωτοβουλία την οποία ανέλαβαν ε, οι αρχές του Κατάρ, οργανώνουν μια τεράστια συγκέντρωση την επόμενη εβδομάδα στο Κατάρ. Θα συμμετέχει μεγάλος αριθμός εκπροσώπων του Εθνικού Συμβουλίου της Συρίας. Μπορεί και πάνω από 400 άτομα. με στόχο να αναδιαρθρώσουν και να ενισχύσουν την εξουσία του Εθνικού Συμβουλίου της Συρίας. Αυτή είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και ελπίζουμε όλοι ότι θα υπάρχει ένα καλό αίσιο αποτέλεσμα, αλλά θα περάσουμε πέρα από το Εθνικό Συμβούλιο στη συγκεκριμένη συγκέντρωση, θα υπάρχουν και εκπρόσωποι άλλων ομάδων ε, της αντιπολίτευσης και εσωτερικής αντιπολίτευσης, θα προσκληθούν όλοι αυτοί για να δουν αν μπορούν από κοινού να συμφωνήσουν ποιο ήταν το πιο βασικό και πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα της Συριακής Αντίστασης ε, ε, και το γεγονός ότι στις αρχές Ιουλίου ε, είχαμε στο Κάιρο την συζήτηση για έναρξη μιας κοινή πλατφόρμας. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει υπάρξει υπόφαση από όλους για συμμετοχή σε αυτή την πλατφόρμα. Θα το θίξουν λοιπόν άλλη μια φορά και θα δουν αν μπορούν να υπάρξει συμφωνία τόσο για την πλατφόρμα όσο και για τη συνέχειά της και να δούμε αν ε, η αντιπολίτευση μπορεί να δημιουργήσει έναν αντιπροσωπευτικό φορέα ο οποίος ε, θα περιλαμβάνει όλους τους ε, συμμετέχοντες στην αντιπολίτευση. Αυτά όλα γίνονται με τον Αραβικό Σύνδεσμο, με τις γειτονικές χώρες οι οποίες έχουν αναλάβει σημαντική ευθύνη για να βοηθήσουν το θέμα της αντιπολίτευσης μέχρι τούδε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της διπλωματίας, και αυτό είναι εξελίξει εδώ και αρκετό καιρό. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να προσεγγίσουμε τα διάφορα μέρη και στα Ηνωμένα Έθνη και αλλού. Ε, ο κύριος Μπραήμι, όπως γνωρίζετε, ήρθε σε επαφή με πολλά, πολλούς από τους ε, διαφορούς συμμετέχοντες. Πήγε και στη Δαμασκό για να συναντήσει τον Μπασάρα Λασάντ. Ε, έχει κάνει αρκετά ταξίδια τον στηρίζουμε και εξετάζουμε με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να μειώσουμε αυτό το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων ομάδων, να δούμε αν μπορεί να υπάρξει κάποια διπλωματική πρωτοβουλία. Ε, η πιο πρόσφατη, ε, οι λεγόμενες συνεδριάσεις ε, του κουαρτέτου με την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία, ε, μέχρι τούδε ήταν ε, τόσο επιτυχές όσο ήλπιζαν οι Αιγυπτιακές αρχές. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν συμμετέχουν μεν σε συνεδρίαση, αλλά έχουν ζητήσει να ενημερώνονται για το τι συμβαίνει και προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί κάποια νέα συνεδρίαση. Εξακολουθώ όμω να αφρονώ ότι πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τον απλό και μόνον λόγο ότι έχει καταφέρει να συγκεντρώσει γύρω από ένα τραπέζι χώρες από την περιοχή που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την παρούσα κατάσταση επιτόπου και επομένως ε, είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία την οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά και επ' αυτού είπα ότι εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, συνεχίζουν και τις επαφές τους με τις Αιγυπτιακές Αρχές. Θα σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Βημό. Δύο ερωτήσει: Καταρχάς, Αναφερθήκατε στις ε, διπλωματικές κινήσεις που έγιναν και τι προβλέπετε να γίνει στις επόμενες εβδομάδες. Ο κύριος Λαυρόμφ ε, το Σαββατοκύριακο νομίζω θα συναντηθεί με την ύπατη εκπρόσωπο. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεάσει και η θέση της Ρωσίας. Και επίσης ε, θα γίνει και μια σημαντική συνεδρίαση στο Μαρακές της ομάδας φίλων της Συρίας, την οποία δεν ξέρω αν αναφέρατε τι άποψη έχετε εσείς για την ε, συνάντηση με τον Λαυρόφ και κυρίως για τη συνάντηση του Μαρακές, γιατί φαίνεται ότι οι Σύριοι δεν είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν στάση. Επίσης, το θέμα των όπλων, το οποίο είναι ιδιαίτερα στη μόδα. Είχαμε και αυτό το αεροπλάνο, το οποίο ξεκίνησε από τη Μόσχα και το σταμάτησαν στην Τουρκία. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα αποδεσμεύτηκε χωρίς ε, ε, τα στοιχεία των πυράβλων που φαίνεται ότι είχε επί του σκάφους. Εμένα αυτή η κατάσταση της Συρίας ε, μου θυμίζει την ταινία του Τσάρλι Βίλσον για το τι συνέβη στο Αφγανιστάν. Μήπως αντιμετωπίζουμε μια αντίστοιχη κατάσταση. Οι Ρώσοι στο Αφγανιστάν είχαν όλη τη στρατιωτική δύναμη και οι επαναστάτες ε, και οι Αφγανοί επειδή δεν είχαν ε, άλλες δυνατότητες δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για την κατάσταση. Θα ήθελα να ξέρω αν εσείς έχετε αντίστοιχη άποψη. Μήπως αλλά Σαντ ε, και ο στρατός του, επειδή παίρνουν όπλα τα οποία έρχονται από το Ιράν ή και το Ιράκ από ό,τι ακούμε, ε, και επειδή οι επαναστάτες από τη Συρία έχουν ελάχιστα όπλα, ε, δεν φαίνεται να μπορεί να κάνει και τίποτα ο ΙΕ, γιατί έχουν ελάχιστα μέσα στη διάθεσή τους. Μήπως βρισκόμαστε ενώπιον μιας πάρα πολύ μεγάλης διένεξης ε, και δεν θα μπορούν οι επαναστάτες να κάνουν τίποτα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα μπορούν να σταματήσουν γιατί θα τους επιτίθεται ο στρατός του, Ασάτ, του Αλασάτ. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Πιστεύετε ότι βρισκόμαστε ενώπιον μεγαλύτερης κρίσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίλαν Μόλαν έδωσε ένα καλό παράδειγμα για δύο λεπτά. Ε, η κυρία Γκόμης. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι στη συγκέντρωση αυτή του Κατάρ, ο κ. Μπραχίμη, ήταν στο επίκεντρο της προσοχής. Εμείς παρακολουθούμε τι συμβαίνει, γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει συνένωση και μεταξύ της αντιπολίτευσης. Και για την ερώτηση του κυρίου Μιλαν και το ρόλο της Ρωσίας και του Ιράν. Εμείς μπορεί να βοηθήσουμε με ανθρωπιστικές κινήσεις ίσως εκτός Συρίας, αλλά έστω σε χώρες που είναι σύμμαχοι στον ΝΑΤΟ, όπως η Τουρκία. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον να προσφέρουμε τα εφόδια που χρειάζονται οι άνθρωποι εντός Συρίας. Ε, δεν μιλάω για ανθρωπιστικούς διαδρόμους στην ίδια τη Συρία. Για γειτονικέ χώρες μιλάω, όπως η Τουρκία η οποία έχει δεχτεί και από, επίθεση από τις δυνάμεις της χώρας, της Συρίας. Έπειτα θα μπορούσαμε να πιέσουμε το Ιράν σε κάποια είδου συζήτηση για τη Συρία. Όχι αναγκαστικά από την πλευρά της Αιγύπτου, αλλά από τη δική μας. Thank you very much, uh, Chairman. ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Βημό για την ε, παρουσίαση αυτή. Μα είπατε τι γίνεται με το Κατάρ, το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία και τι συναντήσει διεθνεί πρωταγωνιστέ. Εγώ θα θέλω να επικεντρωθούμε στο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθεαυτή. Είναι σαφέ ότι είναι πολύ σοβαρά τα θέματα. Στρατηγική ισορροπία και παιχνίδι είναι αυτό που παίζεται μπροστά μα και ε, θα επηρεαστεί η κατάσταση βραχυπρόθεσμα στη Συρία οπωσδήποτε. Οπότε θέλω να ρωτήσω τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει ότι τουλάχιστον θα ενισχύσουμε τι δικέ μα κυρώσει και εμπάργκο. Πολλά ήταν τα παραδείγματα μεταφοράς όπλων από τη Ρωσία στην ε, Συρία μέσω από τα χωρικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τι κάνουμε γι' αυτό. Εσείς τι μπορείτε να κάνετε και τι προτείνετε και στα κράτη-μέλη ώστε να ενισχυθεί και η καταστολή Επίσης, τι πληροφορίες έχετε στην υπηρεσία σας για την ε, ανάδυση των εκτρεμιστικών τάσεων εντός Συρίας όσοι έχουν ε, συνθλιβεί από τη μια μεταξύ της ε, κατασταλτικής κυβέρνησης από τη μια και των ε, δύο εξτρεμιστικών οργανώσεων από την άλλη, που προσπαθούν να αυξήσουν την επιρροή τους. Σε τι θέση βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι δημοκρατικές φωνές, αυτές υπέρ των ανθρωπινών δικαιωμάτων και της ελευθερίας, θα πρέπει να στηριχθούν, να τους βοηθήσουμε. Επίσης μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο την Τουρκία με την τεράστια ροή μεταναστών που δέχεται. Τι είδου συνομιλίε έχουν ξεκινήσει σχετικά και στο επίπεδο του ΝΑΤΟ, αλλά και στο επίπεδο των αυξανόμενων απειλών που αντιμετωπίζει πλέον η Τουρκία. Εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε σε αυτό το τομέα την Τουρκία. Και τι κάνει και με την οικονομική μόχλευση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε υπάρξει ο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο τη Συρία. Αυτό σίγουρα δημιουργεί διάβλου πίεση και άσκηση επιρροή. Εδώ νομίζω δεν έχουμε εκμεταλλευτεί αρκετά τι ευκαιρίε που μας δίνονται και αυτό ίσως να ήταν ένας τρόπος πίεσης εφόσον θέλουμε την πάυση των εχθροπραξιών. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Βήμον, εδώ βρίσκομαι. Ε, η επέμβαση είναι κάτι που μπορεί να σκεφτούμε εφόσον εντείνεται η κατάσταση και ιδίω για τη δημιουργία μια ζώνη απαγόρευση πτήσεων στα σύνορα Τουρκία και Συρία. Και επειδή φαίνεται ότι οι στρατιωτικοί μηχανισμοί τη Συρία είναι ήδη πολύ ισχυροί. Επίση, ισχύουν τα ανθρωπιστικά του διεθνούς δικαίου όπως είδαμε να παραβιάζονται στο κοσυφοπέδιο ή όχι. Τι σχέδια υπάρχουν για τη μαζική έξοδο προσφύγων από την ε, Συρία. Τι πρόβλεψη υπάρχει και θα μπορούσατε να σχολιάσετε επακριβέστερα το ρόλο του Κατάρ που προς στιγμή φαίνεται να χρηματοδοτεί πολλούς και στη Βόρεια Αφρική, τώρα και στην ε, Συρία και ίσως τους πλέον φονταμενταλιστές αλαφίστες που ε, έχουν εξτρεμιστικές τάσεις στη Συρία. Μας ανησυχεί ο ρόλος του Κατάρ και φαίνεται να έχει την τάση να επηρεάζει μαζικά τόσο τη Συρία όσο και τη Λιβύη. Thank you. Κύριε Γενική Γραμματέα, καταρχήν θα ήθελα να σχολιάσω και να σας συγχαρώ εσάς και την ε, Lady Ashton για την στάση σας σχετικά με τη Συρία αλλά ε, γενικώ μας ενδιαφέρει η πολιτική λύση του προβλήματος γι' αυτό και θα ήθελα να γνωρίζω περισσότερα από αυτά τα οποία μας είπατε ήδη μας είπατε πολλά αλλά θα ήθελα να ξέρω πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει περισσότερο στην εξέβρεση μιας πολιτικής λύσης. Γνωρίζουμε τι γίνεται με τους αντάρτες, γνωρίζουμε ποιος θα υπερισχύσει όταν θα τελειώσουν οι χερσαίες μάχες, γνωρίζουμε εάν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η Συρία να γίνει χώρα των Ταλιμπάν, ε, γνωρίζουμε επακριβώς την φύση της διαμάχης στη Συρία. Ξέρουμε ότι η η Συρία και ότι η Τουρκία πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο σαν μια χώρα εμπλεγμένη σε μια διαμάχη αλλά και σε ένα ε, δυνητικά μελλοντικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οπότε θα ήθελα να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που έχετε του θέμα. Thank you, Mr. Thank you very much. Ευχαριστώ είναι προφανές ότι ο Ασάντ θα φύγει μια ώρα αρχίτερα εάν οι τρεις μειονότητες στη Συρία σταματήσουν παθητικά να τον στηρίζουν. Δηλαδή οι ε, χριστιανοί, οι Κούρδοι και οι και μία τρίτη μειονότητα. Υπάρχει ε, αντίθεση στο καθεστώς του Ασάντ και ακόμη και η συνεδρίαση την οποία περιγράψατε στο Κατάρ κύριε Πρέσβη που προσπαθεί να αποδώσει σημασία στο εθνικό Συριανό κίνημα δηλαδή Σουνίτες που είναι ενδεχομένως ένα πρόβλημα για τη Συρία και μπορεί να αποδειχθεί ε, χειρότερο και από το καθεστώς του Προέδρου. Πιστεύω, όπως είπε και ο κύριος Τάνοκ, ότι το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία πρέπει να πιστούν ότι αυτή η μορφή της αντίθεσης ε, θα πρέπει και της αντίστασης θα πρέπει να είναι ένα πιο γενικό σύνολο που θα στείλει ένα μήνυμα εμπιστοσύνης προς όλους τους αντιφρονούντες. Επίσης τελευταίως διάβασα στον τύπο ότι υπάρχει μία προσπάθεια να επιτευχθεί μία προσωρινή κυβέρνηση υπό τον αντιπρόεδρο Φαρού Καλσάρα και αυτό είναι μία προσπάθεια μεταξύ τουρκικού Υπουργού Εξωτερικών και Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών. Υπάρχει ελπίδα για κάτι τέτοιο και ίσως ε, θα είναι η ειρηνική έκβαση της ε, διαμάχης. Επίσης, όταν μιλάμε για πρόσφυγες, και για διάβλους για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πρόσφυγες πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πρόσφυγες δεν πηγαίνουν μόνο στην Τουρκία, στην Ιορδανία, υπάρχουν περισσότερο από ό,τι στην Τουρκία. Και ο, ο, ο, Λίβανος επίσης που αντιμετωπίζει μια επισφαλή ε, κατάσταση εντός των ορίων του. Ο Γενικός Γραμματέας έχει το λόγο. Ευχαριστώ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να, να απαντήσω όσο περισσότερες γίνεται. Πρώτη ερώτηση για τον Υπουργό Εξωτερικών Λαυρόφιεφ. Ναι, έρχεται την Κυριακή Όπως φαντάζεστε με μια διεξοδική ατζέντα για να συζητήσουμε κάποια διμερή στοιχεία που αφορούν τη σχέση μας με την Ρωσία αλλά και για το θέμα της Συρίας. Θα διερευνήσουμε κατά πόσον μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια κοινή συνεννόηση να ακολουθήσουμε τη διπλωματική οδό. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Θα είναι δυσχερή προσπάθεια. Εάν δείτε τι απόσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ των δύο στρατοπέδων, εάν μπορεί κανείς να το ονομάσει έτσι, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μια από τις βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι το θέμα των προϋποθέσεων για την ε, αντιπολίτευση της Συρίας και πολλούς από τους εταίρους μας στη διεθνή κοινότητα, την αντιπολίτευση δηλαδή γενικότερα, οποιοδήποτε, οποιοδήποτε διάλογος σε διπλωματικό επίπεδο μπορεί να ξεκινήσει μόνο με την προϋπόθεση ότι ο Βασίλ Ασάντ θα αφήσει την εξουσία. Θα παρατηθεί. Όμως, αυτό ακριβώς ε, είναι το θέμα. Ο όρος για να υπάρξει μετάβαση να παρατηθεί η κυβέρνηση. Προσπαθούμε να βρούμε κοινό έδαφος μεταξύ των δύο στρατοπέδων και προσπαθούμε να αντλήσουμε διδάγματα και από το παρελθόν και το πώς λύσαμε παρόμοια προβλήματα παλιότερα. Ελπίζουμε να καταλήξουμε σε κάποιο κοινό πεδίο συνεννόησης. που στιγμή δεν έχουμε πετύχει. Έχετε δίκιο και ζητώ συγγνώμη. Ξέχασα να πω ότι η επόμενη συνάντηση των φίλων της Συρίας θα λάβει χώρα στο Μαρακές. Θα προεδρεύσουν οι αρχές του Μαρόκο η οριστική ημερομηνία δεν έχει αποφασιστεί. Λόγος έχει γίνει για την 1η Νοεμβρίου, αλλά θα πρέπει να ενημερώσουμε ξανά μόλις έχουμε πληροφορίες. Πολλά θα εξαρτηθούν από αυτή τη συνάντηση. για το πώς θα μπορούσε να συνασπιστεί η αντιπολίτευση. Θα φανεί αν θα είναι επιτυχής αυτές οι προσπάθειες ή όχι συχνά στη συνάντηση των φίλων της Συρίας. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που προκύπτουν στην ατζέντα είναι η άσκηση πίεσης για να ενωθεί ακριβώς η αντιπολίτευση. Και σε αυτό θα επανέλθω αργότερα. Είναι αρκετά περίπλοκο. Κύριε Μίλανμον, συγκρίνατε την κατάσταση με τι συνέβη στο Αφγανιστάν. Σε ένα βαθμό παρακολούθησα τον παραλληλισμό σα, αλλά εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικό σε τέτοιου είδου συγκρίσει. Είναι πολύ διαφορετικέ Οι καταστάσει. Μιλάμε για ένα πόλεμο του 79-80. Εν τω μεταξύ, μετά από τόσα χρόνια έχουν προκύψει πολλέ νέε τεχνολογικέ εξελίξει. Ό,τι αφορά το εμπάργκο των όπλων, πρέπει να θυμάμαστε πάντοτε δύο πράγματα. Πρώτον, λόγω του αδιεξόδου στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν υπάρχει επίσημο εμπάργκο του διεθνούς κοινότητας. Υπάρχει εμπάργκο των μονομενων κρατών μελών, αυτό που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, και είναι πολύ αυστηρή η εφαρμογή του, αλλά για να απαντήσω και στην τον κύριο Σάκε, στην κυρία Σάκε μάλλον, εδώ έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να πάυσουν τις να εμποδίσουν, να απαγορεύσουν τις πτήσεις ή την, ε, μεταφορά πλοίων. ώστε να ισχύσει πραγματικά το εμπάργκο των όπλων. Αλλά δεν μπορούμε να εμποδίσουμε χώρες που είναι υπέρ του καθεστώτος ε, αντί αυτές που είναι κατά να συνεχίσουν ε, την τροφοδοσία των διαστρατοπέδων με όπλα. Πάντως κάνουμε ό,τι μπορούμε εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο μεμονωμένων κρατών μελών. Είναι αυστηρότατη η εφαρμογή του εμπάργου. Κυρία Γκόμες, ρωτήσατε για τη συνάντηση στην Τόχα και τι γίνεται με τον κύριο Μπραχήμη. Εξ όσων γνωρίζουμε, Η συνάντηση αυτή είχε προκαλέσει και παρανοήσεις και ανησυχίε σε κάποια χρονική στιγμή. Όμως ε, πιστεύουμε ότι ο Αραβικός Σύνδεσμος είναι πλέον θετικός. Η προετοιμασία έχει προχωρήσει πολύ Και ό,τι έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για σχετικά με την επολίτευση έγινε σε στενή συνεργασία με τον Αραβικό Σύνδεσμο. Το παρακολουθούμε πολύ στενά λοιπόν αυτό το θέμα και όλες οι χώρες της περιοχής, όπως η Αίγυπτος και η Λιπή, παρακολουθούν τι συμβαίνει. Επίσης, ευθύ εξ αρχής βρεθήκαμε στην εμπροστοφυλακή προκειμένου να προσεγγίσουμε την αντιπολίτευση και να τους αποστείλουμε σωστά μηνύματα Οργανώνοντα συνομιλίες εδώ στις Βρυξέλλες. Είχαμε συστηματικές λοιπόν επαφές. Ήταν πολύ δύσκολη προσπάθεια, το παραδεχόμαστε, γιατί πραγματικά μεταξύ τους υπάρχουν σοβαρότατες διαφωνίε και διχασμοί και αυτό είναι κατανοητό. Η κατάσταση της κάθε μιας από τις ομάδες αυτές ξεχωριστά είναι ιδιαίτερα δυσχερής και υπάρχει πραγματικά ε, μεγάλη δυσαρέσκεια και απόθεση για τις ε, καχυποψία και δυσπιστία των μεν μεταξύ των δε. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Και σε σχέση με τα όσα συνέβησαν στη Λιβύη, στη Βενγάζη, τουλάχιστον το προσωρινό συμβούλιο μπόρεσε να δημιουργήσει κάποια είδου Στη Συρία δεν το έχουμε πετύχει αυτό ακόμη. Ένα από του λόγου, και συμφωνώ απολύτω με όσα είπε ο κ. Κασουλίδη πριν από λίγα λεπτά, είναι ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Και τους κοινότητες που αναφέρατε, τη χριστιανική, τους Κούρδους, τους Εβραίους, τους Αλαβίτες. Υπάρχει η αίσθηση μεταξύ των κοινοτήτων αυτών ότι είτε ε, με ενεργό ρόλο είτε παθητικά στήριζαν το καθεστώς και παρέμειναν στη θέση αυτή διότι δεν είναι πολύ σίγουροι για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα σε τι θέση θα βρεθεί η κοινότητά τους και αν θα έχει αρκετή προστασία όταν, αν αλλάξουν τα πράγματα. Μία θέση που προσπαθούμε να προωθήσουμε μεταξύ των διαφορών ομάδων της αντιπολίτευσης είναι δείξτε κάποια εμπιστοσύνη μεταξύ σας, κάντε δηλώσεις σχετικά, κάντε κινήσεις και αναλάβετε πρωτοβουλίε, ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία και αυτών των κοινοτήτων. Το μήνυμα αυτό το επαναλαμβάνουμε διαρκώ αλλά θέλει χρόνο. τέθηκε μια ερώτηση για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους εκτός όμως Συρίας και αναφέρατε την Τουρκία. Προσπαθούμε να παράσχουμε μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια καθώς αυξάνει το αριθμό των προσφύγων στην Τουρκία και όπως και εσείς είπατε είναι τεράστιος αυτός ο αριθμός αλλά και άλλοι φτάνουν από την ε, Ιορδανία. Μάλλον και άλλοι έχουν πάει στην Ιορδανία αλλά και στο Λίβανο. Είναι ένα πρόβλημα γενικευμένο. Για την ώρα τα προβλήματά μας με την Τουρκία ήταν κυρίως πρακτικού χαρακτήρα. Οργάνωσαν στα τόπεδα προσφύγων με τρόπο διαφορετικό από το υπόλοιπο Και υπήρξαν παρανοήσεις προκειμένου να φτάσει στο στόχο της η ανθρωπιστική βοήθεια. Νομίζω η κατάσταση θα βελτιωθεί. Καθώς προχωρούμε με τα κονδύλια που θα δώσουμε για την στήριξη των προσφύγων. Νομίζω ότι τα πράγματα θα βελτιώνονται σταθερά. Σε ό,τι αφορά το Ιράν, υπάρχει διχασμός μεταξύ των κατομελών. Κάποιοι πιστεύουν ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή να ζητήσουμε από το Ιράν να λάβει μέρος στις διάφορες συζητήσεις που οργανώνονται στα διάφορα φόρα. Και λόγω βεβαίως και του πυρηνικού προγράμματος και της θέσης του Ιράν σε σχέση με τα πυρηνικά. Πάντω υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι θα πρέπει να λαμβάνουν μέρο λόγω των όσων συμβαίνουν. Η Αίγυπτος προσπάθησε και το συζητούμε αυτό καθημερινά με τους ε, Αιγυπτίους υφήνοντες, αλλά υπάρχει σοβαρή διαφωνία ακόμη μεταξύ των κρατομέλων. Τέχθηκε και μια ερώτηση αλλά νομίζω ότι την απάντησα, για τη βελτίωση της, του πώς υλοποιούνται οι κυρώσεις και πώς επιβάλλονται οι κυρώσεις σε σχέση με τα κράτη-μέλη, συγκρίνοντας τα κράτη-μέλη μεταξύ τους και επίσης για τα εξερευνητικά στοιχεία της αντιπολίτευσης. Εξ όσων ορίζουμε από τις μυστικές μας υπηρεσίες, η αντιπολίτευση που έχει στα χέρια της όπλα είναι μια περίπλοκη περίπτωση. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά στοιχεία. Εξτρεμιστές σαφώς υπάρχουν, διάφορες αντάρτικες ομάδες. Όταν ε, μιλάμε για τον ελεύθερο στρατό της Συρίας, να ξέρουμε ότι πίσω από αυτό το όνομα, το Free Syrian Army, η πραγματικότητα σημαίνει ότι συγκεντρώνονται πολλές αντάρτικες ομάδες, ε, ε ανεξάρτητες σε μια από την άλλη με πολύ ισχυρά τοπικά χαρακτηριστικά που δεν έχουν πολύ σχέση μεταξύ τους. δεν εκπροσωπούν μια γενικότερη τάση στη χώρα. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και ακριβώς λόγω αυτή της πραγματικότητας, όταν μιλάμε για την ανάγκη να προετοιμαστεί η μεταβατική περίοδος, θεωρούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Το να περιμένουμε να εγκαταλείψει την εξουσία το καθεστώς η κυβέρνηση ή να καταρρεύσει και να ελπίζουμε ότι την επόμενη μέρα όλα θα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν και όλα θα μπορούν να προχωρήσουν, αυτό απέχει πόρα από την πραγματικότητα. Εάν δεν ε, προωθήσουμε τώρα τη διπλωματική διαδικασία προτού συμβούν όλα αυτά, η αντιπολίτευση εντός και εκτός της χώρας Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι θα πρέπει να προετοιμαστεί για να συζητήσει. Πρέπει να εργαστούμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση και για την ε, επόμενη μέρα θα είναι πολύ σημαντικό να ασκηθεί πίεση μέσω του εμπορικού, των εμπορικών μας σχέσεων. Ακόμη και η συνεργασία μας, ε, βεβαίως ήταν ε, ένας σημαντικός εταίρος για την Ευρώπη η Συρία. Αυτό είναι ατού στα χέρια μας προκειμένου να μπορέσουμε στο μέλλον να συνεργαστούμε με τις νέες αρχές της Συρίας μόλις προκύψουν. Κύριε Τάνοκ, ρωτήσατε κάτι για μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και γενικότερα για το ζήτημα της στρατιωτικής παρέμβασης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καλώς μας θυμήσατε ότι για στρατιωτικές επιχειρήσεις χρειάζεται και η στήριξη του ΟΗΕ και κάποιο ψήφισμα του ΟΗΕ. Αλλά εάν δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε τέτοιο ψήφισμα στα χέρια μας, είδαμε, όπως στην περίπτωση του Κωσυφοπεδίου που και ο ίδιος αναφέρατε, είδαμε κάποιοι εταίροι της διεθνούς κοινότητας να προχωρούν παρά την απουσία ψηφίσματος. Η δυσκολία εδώ είναι ότι αν θέλουμε να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, η στρατιωτική επιχείρηση που θα αναγκαζόμασταν να σχεδιάσουμε, είτε για ανθρωπιστικού διαδρόμου, είτε για μια ζώνη αναχέτηση, είτε για μια ζώνη απαγορεύση πτήσεων, οποιαδήποτε τέτοια ζώνη θέλαμε να δημιουργήσουμε, θα απαιτούσε στρατιωτική στήριξη. Λόγω των δυνατοτήτων του στρατού της Συρίας, επειδή έχουν τέτοιε δυνατότητες άμυνα, έχουν ε, πάρα πολύ μεγάλο αεροπορικό ε, αεροπορική δύναμη, ελικόπτερα, θα πρέπει να προετοιμαστούμε πολύ καλά. Δεν θα έχει καμία σχέση με το τι έγινε στη Λιβύη. Και οι χώρες που θα λάβουν μέρος, χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες και άλλοι, το σκέφτονται, το σκέφτονται δυο φορές πριν πάρουν κάποια απόφαση. Τι παιχνίδι παίζει το Κατάρ τώρα. Εξ όσων φαίνονται, σίγουρα είναι υπέρ της μιας πλευράς και είδαμε από τη συνάντηση στην Τόχα ότι προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των διαφορών ομάδων της αντιπολίτευσης. Το Κατάρος τώρα στήριζε κυρίως το Εθνικό Συμβούλιο της Συρίας. Τώρα όμως με τη συνάντηση που την στην Τόχα προσπαθούν να ανοίξουν κάπως το πεδίο και να συμπεριλάβουν περισσότερους. Συγκεράζοντας και άλλα στοιχεία της αντιπολίτευσης. Το αν θα πετύχουν ή όχι είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε, αλλά θα τους παρακολουθούμε στενά. Τέλος, και πολύ σύντομα, για να απαντήσω και σε άλλες ερωτήσεις που τέθηκαν και δεν πρόλαβα να απαντήσω για την ενδιάμεση κυβέρνηση. Η ιδέα αυτή έχει συζητηθεί. Θα το ξανακούσετε μάλλον και με τη συνάντηση της Δόχα. Τώρα, αν ο Φαρούκαλ ε, Σαχάρ πρέπει να ηγηθεί ή όχι, ή κάποιος άλλος, είναι κάτι που θα μας απασχολήσει, γιατί υπάρχουν προσωπικότητες που έχουν συνεργαστεί με το καθεστώς επί χρόνια και βεβαίως στην αντιπολίτευση υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα ως προς τις συγκεκριμένες προσωπικότητες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Εάν επιτρέψετε, θα έχουμε ακόμη τέσσερις ερωτήσεις, ενός λεπτού η καθεμία. Ο κύριος Αγκουράκης πρώτος, μετά ο κύριος Αλαβράκος, ο κύριος Κράισελ Ντόρφελ και ο κύριος Βότσον. Ο κύριος Αγκουράκης έχει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να επισημάνω ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή μεγάλης κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης και της επέμβασης ξένων δυνάμεων στη Συρία. Και μου κάνει εντύπωση που ε, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης δεν ανισχύει γι' αυτό. Ε, τα επεισόδια στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας ε, και ο τρόπος που αντέδρασε το ΝΑΤΟ δείχνουν ότι μπορούμε να περιμένουμε ακόμα χειρότερα πράγματα στο άμεσο μέλλον. Επίσης το επεισόδιο με το αεροπλάνο στην ε, Τουρκία είναι τελείως απαράδεκτο. Ο ίδιος είπατε ότι δεν υπάρχει εμπάργκο πωλήσεων όπλων, άρα η ενέργεια των τουρκικών αρχών ήταν τελείως παράνομη και θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Μάλλον θα κάνει τίποτα γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θέλετε ως υπηρεσία εξωτερικής δράσης όσο πιο γρήγορα γίνεται να υπάρχει μια κλιμακούμενη ξένη επέμβαση στη Συρία γιατί δεν μπορείτε αλλιώς να λέξετε την ε, κατάσταση. Αυτό που θα ήθελα εγώ να σημειώσω είναι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή επέμβαση του ΝΑΤΟ ε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή ε, μια κυβέρνηση με ξένε δυνάμει και με ξένα δεκανίκια στη Συρία γιατί θα έχει το ίδιο μέλλον όπω και αυτή του Αφγανιστάν. Ευχαριστώ κύριε Thank Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε. Πρόεδρε. Ε, θεωρώ πολύ ικανοποιητική την έμφαση που δίδεται στην ανθρωπιστική βοήθεια των πληθυσμών στη Συρία. Συνάμα όμως θεωρώ επικίνδυνη την έμεση απειλή του Συριακού καθεστώτος σχετικά με τη χρησιμοποίηση χημικών όπλων έστω και αν αυτό εμφανίζεται ότι θα γίνει σε περίπτωση ε, ξένης επέμβασης. Σύμφωνα με πολλούς Αναλύτε σε μια εμφύλια σύλληξη όπω συμβαίνει τώρα, το πιο πιθανό σενάριο είναι τα όπλα να περιέχουν στην κατοχή των ανταρτών ή και ομάδων όπως η και ομαδων οπω η Χεσμολάχ ή η Αλκάιντα. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον ε, κύριο Γενικό Διευθυντή να μας ενημερώσει προς ποια κατεύθυνση έχει κινηθεί η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ως προς αυτό το ζήτημα ή αν έχει πληροφορίες ε, σχετικά με κινήσεις άλλης ε, ε, ομάδος ή δυνάμεως από τη διεθνή κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μαζί με την ε, Κάτι Άστον ο κύριος Βιλμό μας παρουσίασε μια πολύ σαφή εικόνα για το τι γίνεται στη Συρία τι γίνεται όμως στην Ιορδανία διότι εκεί δεν έχουν επιληθεί τα θέματα της Παλαιστίνης και επιπλέον η Συρία, ο Λίβανος όλα αυτά φορτώνει ακόμη περισσότερο την εικόνα πώς αξιολογεί ε, η υπηρεσία στην κατάσταση στην Ιορδανία, ο Σερ Γκράχαμ Βότσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο ε, Βήμο εάν ε, μετά την ε, αποτυχία της συναντήσεως στο Κάιρο τον Ιούλιο και της επερχόμενης συναντήσεως την επόμενη εβδομάδα στο Κατάρ εάν πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει ένα πολιτικό μέλλον για τη χώρα αυτή και σχετικά με τις Ηνωμένε Πολιτείες έχει γίνει μια συζήτηση για την κατάρτιση μιας task force στην Ιορδανία και θα αποδώσει. Επίσης το αεροπλάνο που έφυγε από την Ρωσία ε, για να πάει στη Συρία ε, παραβίαζε τους κανόνες πολιτικής αεροπορίας σχετικά με το φορτίο το οποίο μετέφερε. Πολύ λοιπόν. σύντομα για την ε, πρώτη ερώτηση. Πραγματικά εμεί ανησυχούμε ιδιαίτερα για αυτό που συμβαίνει. Νομίζω ότι είπα ότι η εκπροσωπο σας εξήγησε πριν από δύο ημέρες ε, πόσε επαφές έκανε την ε, εβδομάδα που ήταν στη Νέα Υόρκη με όλες τις πλευρές προκειμένου να προσπαθήσει να πιέσει ε, την πολιτική κατάσταση μέχρι του σημείου που μας επέκριναν ότι είμαστε πολύ αφελείς. Το να λέμε ότι αδρανούμε λοιπόν ότι, και ότι θα κάνουμε, πρέπει να κάνουμε περισσότερο δεν είναι σωστή αξιολόγηση της κατάστασης. Κάνουμε πολλά όπου μπορούμε σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας, προσπαθούμε να πιέσουμε την αντιπολίτευση προς περισσότερη ενότητα και προσπαθούμε όλες οι ομάδες να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πάλι και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και με τον Σεργέη Λαυρόφ ε, την Κυριακή. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ρεαλιστέ. Δεν θα είναι εύκολη κατάσταση, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να πιέσουμε κι άλλο και να συνεχίσουμε. Όσον αφορά τα χημικά όπλα τώρα, εν συντομία, είμαστε σε επαφή με όσους έχουν πληροφορίες από αυτού του ζητήματος. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αν μας ζητηθεί με τις δικές μας τις δυνατότητες, αλλά προς το παρόν ε, αυτό που κάνουμε είναι να παρακολουθούμε στενά ε, πού μπορεί να βρίσκονται αυτά τα τόσο επικίνδυνα όπλα και αν έχουν μεταφερθεί ε, σε κάποια άλλη τοποθεσία. Ε, κάτι για την Παλαιστίνη. Οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες, μεταξύ άλλων, θα έπρεπε να το είχα αναφέρει και νωρίτερα. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, διότι σε πολλές από αυτές τις χώρες που είναι κοντά στη Συρία ε, υπήρχαν Παλαιστίνοι ε, πρόσφυγες κοντά στα σύνορα και ε, τώρα χρειάστηκε να μεταφερθούν. Και μέρος της ανθρωπιστικής μας βοήθειας αφορά ε, ακριβώς αυτό το πρόβλημα των Παλαιστινίων προσφύγων, που νομίζω ότι αρχίζει να γίνεται όλο και πιο ανησυχητικό. Θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε στενά. Τέλος, για τις ερωτήσεις ε, που έθεσε ο κύριος Βότσον, η πλατφόρμα του Καΐρου εξακολουθεί να υπάρχει. Έχει αποτύχει βέβαια προς το παρόν ε, και δεν την υποστηρίζουν όλοι, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Και ζητήσαμε από τις αρχές του Κατάρ μήπως θα μπορούσε να αποτελέσει και βάση συζήτησης μεταξύ των διαφόρων ε, ε, μελών της αντιπολίτευσης στην Τόχα από την επόμενη εβδομάδα και μετά και η απάντηση ήταν καταφατική. Είναι ακόμα λοιπόν στο προσκήνιο σε πολιτικό επίπεδο. Όσον αφορά την Task Force των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να την απευθύνεται ε, την ερώτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι σε μένα. Γνωρίζουμε όλοι ότι στην Ιορδανία όλοι μας και οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ιδιαίτερα τις αρχές τη Ιορδανία που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στα σύνορά του και θα συνεχίσουν. Όσον αφορά τη ρωσική πλευρά, δεν ξέρω αν θα. και το αεροπλάνο αυτό, δεν ξέρω αν θα τεθεί το ζήτημα αυτό, αν θα το θίξει κάποιο. Αλλά νομίζω ότι από εδώ και στο εξή, μέχρι την Κυριακή, θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά για να δούμε αν υπάρξει οποιαδήποτε δήλωση από τη Μόσχα για το θέμα. Θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Το ότι ήρθε σήμερα εδώ ο Γενικός Γραμματέας είναι κάτι το οποίο αιτιολογεί την καθυστέρηση της ψηφοφορίας διότι εφόσον αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν νομίζω ότι είναι ένα επιχείρημα και γι' αυτό και δικαιολογώ αυτούς οι οποίοι καθυστέρησαν να έρθουν. Κυρίες και κύριοι, ας ξεκινήσουμε τώρα το σημείο 14. η σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με τη νέα συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, Ρωσίας. Ο κύριος Σουόμποτα, εισηγητής, ε, δεν θέλει να παρέμβει και προχωράμε κατευθείαν στην ε, ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ της πρώτης συμβιβαστικής τροπολογίας. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην τροπολογία 62. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ Μα το καλύψαμε. Το 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ε, συγχαίρω την ε, ετούσα την τροπολογία και τον τροπολογόντα, δηλαδή εμένα. Το 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ το 73 και το 72 έχουν καταργηθεί Οπότε είμαστε τώρα στο 76. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. 76. Λίγη. Εγκρίθηκε 30 υπέρ 22 κατά. Ε, δεύτερη συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ερχόμαστε τώρα στην 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στο 91 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος Παρακαλώ να συμμετέχετε στις ψηφοφορίες, οι 125. Λίγοι. Απερίφθη. 37 κατά, 17 υπέρ. 126 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 127 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 128 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 132 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 133 χρωριστή ψηφοφορία σε τρία τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο, ελέγχουμε το δεύτερο μέρος και ε, λίγη ψηφοφορία 27 ε, υπέρ, 28 κακά. Ε, δεν χρειάζεται βέβαια κατόπιν αυτού να ψηφίσουμε για τον όρο ε, real, real, πραγματικό διότι εδώ η πραγματικότητα έχει γίνει εξωπραγματικό στην θέση αυτή. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 σε δύο τμήματα το πρώτο τμήμα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, περίφθη Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ερχόμαστε στο 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 σε δύο τμήματα το πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 171 σε δύο τμήματα ποιος είναι για το πρώτο τμήμα υπέρ του πρώτου τμήματος κατά ε, ε, ε, ενεκρίθη δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο μέρος της 171 λίγη υπερψηφίστηκε με 28 υπέρ 27 κατά 172 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 174 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 175 σε τρία τμήματα για το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 178 υπέρ, Το 177 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάθονται με στην αίθουσα αλλά δεν ψηφίζουν λέει ο πρόεδρος. 39 υπέρ και 16 κατά. Ποιος ζήτησε να ελεγχθεί. Η κυρία Μουνής. Εκατόν εξήντα οκτώ υπέρ. 178 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. 180 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι για το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος. Λίγη. Ενεκρίθη. Το δεύτερο τμήμα έχει καλυφθεί από τη συμβιβαστική 10. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 182 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 183 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 184 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 185 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος Λίγη ψηφοφορία. Ενεκρίθη 29 υπέρ, 25 κατά. 186 υπέρ, κατά, αποχές, ενεκρίθη. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, ενεκρίθη. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λίγη. 30 υπέρ και 24 κατά. Το 13 καταπίπτει και ψηφίζουμε την τροπολογία 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 15 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 16 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 17 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 18 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 19 υπέρ κατά αποχές απερίφθη από το 20 έως το 24 μπορούμε να ψηφίσουμε σε μία δόση ποιος είναι υπέρ όχι δεν θέλετε ένα ένα 20 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 21 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 22 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 23 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 24 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 25 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη Συμβιβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, ενεκρίθη. Τώρα ερχόμαστε στην 33 υπέρ, κατά, αποχές, ενε, απερίφθη. 34 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 35 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Συμβιβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, ενεκρίθη. 36 υπέρ, μάλλον 41 41 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 42 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 44 σε 4 τμήματα πρώτο τμήμα εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ 49 ηλεκτρονικός έλεγχος λίγη με 35 υπέρ και 18 κατά κυρία Γκομές, την τρίτη φορά θα πιούμε σαμπάνια. Ρώσικη σαμπάνια. 50 υπέρ κατά αποχές επανερχόμαστε στην 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε «51 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος» κατά αποχές εγκρίθηκε. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά ε, ε, απερίφθη. 2 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. 3 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη ηλεκτρονική ψηφοφορία του συνολικού κειμένου. Λίγοι. Η έκθεση ψηφίστηκε με 53 ψήφους υπέρ, μία αρνητική και μία αποχή αλλά συγχαίρουμε τον ε, κύριο Σόμποντα. Νομίζω ότι ήταν μια ισχυρή ε, κίνηση για ένα τέτοιο, μια τέτοια έκθεση ότι υπήρξε τόσο ευρία συνένεση στην έκθεση αυτή. Θα χρειαστεί χρόνο για να συνέλθει ο εισηγητής. Τώρα ερχόμαστε στο σημείο 15 Καζακστάν, η κυρία Γιακονσάρη. Ε, θέλετε μήπως να παρέμβετε, αν όχι ερχόμαστε στην τροπολογία 39. Υπέρ, κατά. Αποχές, απερίφθη. Συμβιβαστική 8, υπέρ, κατά. Αποχές, ενεκρίθη. Ε, τροπολογία 42, υπέρ, κατά. Αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ε, αν όλοι ψήφιζαν δεν θα χρειαζόντουσαν τόση ηλεκτρονική έλεγχη. Λίγοι. 28 υπέρ, 22 κατά, είναι κρίθη. 43 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 44 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. Ερχόμαστε τώρα στις 46 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. 51 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. 52 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 53 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 55 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 57 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 58 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 59 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 60 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη ερχόμαστε στην 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και φτάνουμε στην 66 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι για το, υπέρ του πρώτου τμήματος, τρία τμήματα μάλλον, ε, υπέρ κατά αποχές. Ενεκρίθη. Η κυρία Γέγκλε πρέπει να μας λέει και προφορικά τι θα κάνουμε. Ποιος είναι υπέρ του δεύτερου μέρους. Υπέρ κατά. Νομίζω ότι ενεκρίθη. Τρίτο τμήμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 66. Λίγοι. Ενεκρίθη. Τρίτο τμήμα. Λίζαμπετ, για πρόσεχη γιατί σε λιγάκι θα μου αγοράσει και εμένα σαμπάνια να με κεράσεις. Ποιος είναι υπέρ του τρίτου τμήματος, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην 67, υπέρ κατά απόχέ. απορρίπτεται. 68, υπέρ κατά απόχέ. εγκρίθηκε. 70, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 71 ενεκρίθη 27 υπέρ 23 κατά 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 72 υπέρ είναι η ίδια πλειοψηφία όπως και πριν ξαναψηφίζουμε ηλεκτρονικά το 71 71 λίγη 28 υπέρ, 22 κατά. «72». Μέχρι το μεσημέρι θα έχω μεθύσει από τις σαμπάνιες που κέρδισα στα στοιχήματα. 72 υπέρ, μεθυσει απο τους σαμπανιες Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και ερχόμαστε στην 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και πάλι. Νομίζω ότι είναι λίγο πολύ ίδια πλειοψηφία. Λίγη. 28 υπέρ 21 κατά ενεκρίθη 78 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 81 και 102 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 82 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος Λίγη. Ενεκρίθη 29 υπέρ, 21 κατά, πάντοτε ίδια πλειοψηφία, 83 ε, υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 84 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. 87 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. 88 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 89 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 90 ε, πρέπει να συμπεριλάβουμε και τον όρο social του εισηγητή υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90... για το 94 ηλεκτρονικός έλεγχος εμένα μου φάνηκε ότι είχε υιοθετηθεί αλλά ας το δούμε ορισμένοι έχουν ξεχάσει τις κάρτες τους λίγοι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 Λίγη η ψηφοφορία. Απερίφθη με 27 κατά και 21 κατά. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές ενεκρίθη. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές ενεκρίθη. 113 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 114 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 115 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 116 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη ε, τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 10 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 11 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 12 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 13 υπέρ έλεγχος για τη 12 Όπως ξέρετε ότι το αντικείμενο και η πλειοψηφία δεν επικαλύπτονται πάντοτε. Λίγοι. 27 υπέρ, 23 κατά. 13 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 καταπίπτει. 15 και 17 είναι ταυτόσημα συν προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αυτό πρέπει να το ελέγξουμε δεν μπορεί να είναι διαφορετικά ξεκινάει η ψηφοφορία λίγη απερίφθη 38 κατά 12 υπέρ συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε ερχόμαστε στην τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές ε, νεκρίθη Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. Και τώρα ερχόμαστε στην 28 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. 32 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. 35 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Λίγη ψηφοφορία. 26 υπέρ και 25 κατά ενεκρίθη. 36 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι για το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι για το δεύτερο. Μάλλον ποιος είναι κατά. Αποχές ενεκρίθη. Δεύτερο τμήμα. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος έληξε απερίφθη 24 υπέρ 26 κατά ε, τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές πάλι η ίδια πλειοψηφία τέσσερα. υπέρ κατά ενεκρίθη είναι τα ένα πρέπει να δουλέψουμε λίγο γιατί εν μέρη αυτό έχει καλευθεί και θα πρέπει να υπάρξει κάποια επεξεργασία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Οπότε δεν χρειάζεται καν να το επεξεργαστούμε. Είναι τα δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Είναι τα πέντε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ίντα 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ίντα 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ίντα 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ίντα 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ίντα 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για να κάνουμε έναν έλεγχο. Λίγοι. 25 υπέρ, 24 κατά και μία αποχή. Είναι τα 11. Υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Είναι τα 12. Υπέρ, κατά, αποχές, κρίθη, Είναι τα 13. Υπέρ, κατά, αποχές, ενεκρίθη. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη συνολική έκθεση ξεκινά. Λίγη. Ενεκρίθη με 43 υπέρ, καμία αρνητική και μία ε, επιφύλαξη. Τι θα γίνει, θα έχουμε επεξηγήσεις ψήφου, ρωτάει ο κύριος Πάσκα. Τώρα όμως πρέπει να κάνουμε γρήγορα διότι στις 11 έχουμε ε, την ε, ακρόαση και θα μας ενημερώσει ο κύριος ε, Μιλάν Γκάμπροχ σχετικά με την αποστολή εκλογικών παρατηρητικών στις κοινοβουλευτικές εκλογές στη Γεωργία την 1η Οκτωβρίου 2012. Ε, πέραν αυτού ο κύριος Ντοζό Μπαζέσκου, η κυρία Νικολάη Ταράντ, νικολαη ταραντ η μπραζας και ο κύριος Πίκολα.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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτές. Για μένα είναι μεγάλη τιμή που έχω την δυνατότητα σαν Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας για την επίβλεψη των βουλευτικών εκλογών ε, στη Γεωργία ε, να μπορέσω να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της ε, αποστολής μας σε συνεργασία συνεργασία με την ε, Κοινοβουλευτική Συνέλευση και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ. Ε, καταφέραμε να καταρτήσουμε μία κοινή ε, τοποθέτηση και ήμασταν λίγες μέρες πριν τις εκλογές στην Γεωργία και είχαμε ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αποστολής του κυρίου Νικολάη προηγουμένως σχετικά με την κατάσταση λοιπόν της γεωργίας ήμασταν πολύ ενήμεροι και σχετικά με την εκπροσώπηση των μέσων ενημέρωσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Παρακολουθήσαμε την εκλογική διαδικασία στη γεωργία καθώς επίσης και ε, την προετοιμασία των εκλογών και την αξιολογήσαμε ε, υπήρχε το δικαίωμα ε, ελευθέρης εκφράσεως λόγου και ε, ελευθέρας συγκεντρώσεως, ελευθερία συγκεντρώσεων ε, χαρακτηρίστηκε λοιπόν η προεκλογική περίοδος από αυτό, αυτή την ατμόσφαιρα και δεν υπήρξαν ε, αρνητικές εκδηλώσεις. Οι πολίτες ήταν υπέρ ε, των εκλογών. Προηγουμένως υπήρχαν εντάσεις και φόβοι για εκδηλώσεις βίας για τη νύχτα με μετά τις εκλογές, πράγμα όμως το οποίο ευτυχώς δεν υλοποιήθηκε και χθες είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όλη την διεξαγωγή ε, και είδαμε ότι στην Τυφλίδα, στο καφέ κλικ είδαμε ότι οι κανόνες είχαν γίνει σεβαστές και σε ορισμένα εκλογικά τμήματα υπήρχαν λάθη. Είδαμε όμως και, ε, και ε, εκλογής που περίμεναν να εξασκήσουν το δικαίωμά τους χωρίς όμως να υπάρχουν παράνομες κινήσεις και η Κεντρική Επιτροπή ε, μας κοινοποίησε τα αποτελέσματα τη Δευτέρα και 40,3% καλύφθηκαν από το Εθνικιστικό Κόμμα και 43% από τους ε, ισχύσαντες. Το νέο κοινοβούλιο εκπροσωπείται τώρα από αυτές τις δύο ομάδες πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι το ε, κυβερνητικό κόμμα από τη άλλη μεριά και η αντιπολίτευσης συμμετείχαν υπήρχαν ορισμένα παράπονα σχετικά με την ε, διαδικασία και τη διεξαγωγή των ε, ε, εκλογών ανακοινώθηκε από τον κύριο Σακασβίλη ότι παραδέχεται το αποτέλεσμα των εκλογών και θα υπάρξει πολιτική ρύθμιση οποία είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων στη Γεωργία. Τέλος θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία στη Γεωργία τα τελευταία χρόνια έχει ε, προχωρήσει πολύ. Οι πολίτες της Γεωργίας έχουν ε, βασικά δικαιώματα και ε, θεμελιώδεις ελευθερίες και για πρώτη φορά υπήρξαν δημοκρατικές εκλογές στην η Γεωργία που αποφάσισαν την αλλαγή ε, της κυβέρνησης και η κυβέρνηση παρεδέχθη την ήττα της η Γεωργία έχει προχωρήσει στην συνεργασία με την Ευρώπη και όσον αφορά το δικαίωμα του συνέρχεστε ε, σας έχω ήδη ενημερώσει τώρα σχετικά όμως ε, με την προσχώρηση του ΠΟΕ, στον ΠΟΕ ε, φαντάζομαι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καλέσει την Γεωργία για να από προωθήσει την ε, ε, συνεργασία και θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την βοήθειά τους. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε ε, και θέλω να ευχαριστήσω και τους συμμετέχοντας στην αποστολή ως παρατηρητές για τις εκλογές παρόλες τις ατέλειες τις οποίες συζητήσαμε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία ελεύθερη κατάσταση, υπήρξαν ορισμένες εντάσεις ε, και γι' αυτό η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή κινήθηκε επαγγελματικά. Εγώ είχα υπάρξει προ δύο ετών παρατηρητής για τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχαμε αντιληφθεί ότι βαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση και βλέπω ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί βελτιωθεί. Πράγμα το οποίο ε, θεωρώ ότι ε, εγώ έχασα λόγω επιφυλάξεων, κέρδισε όμως η δημοκρατία, ήταν μια σημαντική στιγμή για την δημοκρατία και αυτή η ειρηνική εξέλιξη ελπίζω ότι θα συνεχιστεί και θα μπορέσουμε στις επόμενες εκλογές να έχουμε πάλι προϋποθέσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε μία ειρηνική μεταφορά της εξουσίας πράγμα που θα είναι ένα ευίωνο μήνυμα από την Γεωργία και θα αποτελέσει και ένα βασικό μήνυμα για άλλες χώρες της περιοχής κατά τρόπον ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ε, προοπτική αυτών των χωρών. Επίσης ελπίζω ότι το γεγονός ότι η χώρα πρέπει να προσβλέπει προς την ε, ε, Δύση δεν περιελήφθημένες ε, στα σχόλια του Υπουργού Εξωτερικών αλλά ελπίζω ότι αντιμετωπίζει, συμφωνούν με το πνεύμα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας να ευχαριστήσω και εγώ τον επικεφαλής της αποστολής και νομίζω ότι η αποστολή έκανε πολύ σωστή δουλειά όσον αφορά τη διεξαγωγή των εκλογών και την κατάσταση μετά τις εκλογές συμφωνώ πλήρως με τον κύριο Μπρόκ η πρώτη φορά στην ιστορία της σύγχρονης γεωργίας όπου υπάρχει μία ειρηνική αλλαγή στην εξουσία και η γεωργία έχει καλύψει μία από τις προϋποθέσεις της δημοκρατίας, δηλαδή ε, μία εναλλαγή και ε, ε, αλλαγή της κυβέρνησης. Νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε την γεωργία να εξελιχθεί και θα κάνουμε έκκληση και προς τις δύο πλευρές και τους κερδισμένους και τους χαμένους και θα τους ζητήσουμε να συνεργαστούν προς όφελο όφελος της ε, εξελίξεως στη χώρα και προς όφελος των αλλαγών που πρέπει να εφαρμοστούν για να προοδεύσει η χώρα και στο πνεύμα των ε, διατλαντικών δομών είτε ε, της του ΝΑΤΟ είτε τη ΣΧΙΑ, ε, δηλαδή της οργανώσεως που προωθεί την ε, συνεργασία στην περιοχή. Ε, έχω να κάνω ακόμη ένα σχόλιο σχετικά με την επόμενη αντιπροσωπεία παρατηρητών. Ε, έχω συναντήσει ορισμένους από τους αντιπροσώπους και αντιλαμβάνομαι ότι αυτοί δημοσίευσαν χωριστά την ενημέρωση προς τον τύπο και πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος των δηλώσεων προς τον τύπο δεν πρέπει να γίνεται έτσι δηλαδή χωριστά ας συνεννοηθούμε πρώτα μεταξύ μας και μετά αφού συνεννοηθούμε θα έπρεπε να εκφράσουμε μία ενιαία ε, παρουσίαση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζάιρος Βόλσκι. Ευχαριστούμε για την εισήγησή σας. και είναι καλό που οι εκλογές εξελίχθηκαν με θετικό τρόπο. Είναι σαν μια αναδρομική, μια πύριος νίκη του κυρίου Σακασβέλη, ο οποίος βγήκε από τις εκλογές. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όρος για τις εκλογικές αναμετρήσεις είναι η διαφάνεια και περιορισμένη χρήση κοντιλίων για τη χρηματοδότηση. Μπορούν ε, οι διαγωνιζόμενοι να χρησιμοποιήσουν χρηματοδότηση, αλλά υπάρχουν όρια. Και πάντοτε με διαφανείς διαδικασίες και με κάποια περιορισμούς, όπως είπα. Αυτό είναι το σύστημα στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις εκλογές της Γεωργίας ένα τεράστιο ποσό χρημάτων, 300 εκατομμύρια δολάρια εκτιμάται, χρησιμοποιήθηκαν από το κόμμα του Γιάννασβίλη. Οι παρατηρητές το έλαβαν αυτό υπόψη, είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Ε, το συμπεριέλαβαν στην αποτίμησή τους για το κατά πόσο ήταν νόμιμες εκλογές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Κάμπερνοχ για, την ομάδα των παρατηρητών για το έργο τους και για την εισήγηση σήμερα. Θα μπορούσε να μας δώσει κάποια συμβουλή για το τι θα έπρεπε να γίνει στο μέλλον ώστε τα κόμματα στην Γεωργία να συγκεντρωθούν και να συμφωνήσουν για τους κανόνες των προεκλογικών εκστρατιών, διότι συμφωνώ με την άποψη των παρατηρητών το αποτέλεσμα ήταν ε, δίκαιο και νόμιμο, όμω, κάποιε πτυχές ε, της προεκλογική περίοδου που να μην, ίσως να μην είδαμε και επαρκώς όλοι μας ήταν σημαντικές. Εκφοβισμός ε, υπήρξε, κάποιοι από τους υποψηφίους δέχτηκαν πιέσεις Ο κύριο Κάμπερνοχ λοιπόν οι συναδελφοί του έχουν ε, άποψη για το πώ θα μπορούσαμε στο μέλλον να επηρεάσουμε τη διαμόρφωση των κανόνων και να λειτουργούν ακόμη πιο εύρυθμα τα συστήματα. Νομίζω η δημοκρατία όπω έλεγε και ο Τσέρτσιλ είναι ένα κακό σύστημα. Είναι όμω καλύτερα από οποιαδήποτε εναλλακτική. Πάντω σίγουρα πολλά μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η λειτουργία του. Και νομίζω ότι η δέσμευση της Ευρωπαϊκή Ένωσης μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους οργανισμούς ώστε να διασφαλίσουμε ότι ε, συνεχίζει να επιτελεί πρόοδο η λειτουργία της δημοκρατίας σε χώρες όπως η Γεωργία είναι κάτι το ευκταίο. Ευχαριστούμε κυρία Νίκολαη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμμετείχα σε αυτή την αποστολή και θεωρώ ότι οι εκλογές ήταν πραγματικά ανταγωνιστικές και ελεύθερες και δίκαιες. Βεβαίως κάποια μικροπεριστατικά υπήρξαν. Όμως αυτό είναι μάλλον σύνηθες. Η προεκλογική εκστρατεία είχε κάποια μικραβία επεισόδια, κάποιες κινήσεις της κυβέρνησης, όμως τελικά αυτό δεν μέτρησε στο κλικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η πόλωση σε δύο βασικά κόμματα θα είναι επίτευμα για την ε, δημοκρατία στη Γεωργία και Νομίζω ότι θα μπορούσαμε και εμείς να βοηθήσουμε στη σύνταξη κανόνων ενός καταστατικού για τις προεκλογικές εκστρατείες. Ε, θα... Ήταν καλό να συμμετέχουμε στην προσπάθεια σταθεροποίηση αυτού του νέου δημοκρατικού καθεστώτο. Πάντω η Γεωργία παραμένει μια δημοκρατική χώρα και συνεχίζει να συμμερίζεται τι αξίε μα. Ευχαριστούμε κυρία Λούνατσεκ. Κυρία Λούνατσεκ, μην με κοιτάτε τόσο λυπημένη. Δεν είμαι λυπημένη. Ευχαριστώ και από πλευράς μου ε, τον συνάδελφο για την έκθεση και την εκτίμησή μου θα ήθελα να εκφράσω γιατί κάνατε αυτή την παρατήρηση των εκλογών. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, αποτελεί καλή ένδειξη για τη δημοκρατία στη Γεωργία, ιδίως μετά την πόλωση την οποία διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Εν τέλει θεωρώ ότι τη νίκη την είχαν οι πολίτες της Γεωργίας ε, με τον τρόπο που διεξήχθησαν οι εκλογές παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες ελλείψεις και κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να βελτιωθούν στο μέλλον. Από γεωπολιτική σκοπιά ε, και το ρόλο που θέλει να διαδραματίσει η Ρωσία στον τομέα είναι πολύ σημαντική η νίκη, διότι μια πραγματικά δημοκρατική γεωργία για τον Πούτιν και τους φίλους του είναι πραγματικά πρόβλημα, θα τολμούσα να πω. Δεν θα τους άρεσε καθόλου. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθησαν οι εκλογές και το τελικό αποτέλεσμα ήταν πολύ σημαντικό. Δύο ερωτήσεις προς τον συνάδελφο. Ε, κάποιος άλλος αναφέρθηκε και πάλι στη χρηματοδότηση των κομμάτων. Ε, τι διαπιστώσατε, υπήρχαν κάποιες επικρίσεις από πλευρά σας για το θέμα αυτό. Και επίσης, υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί που δεν είναι ισχυρισμοί, είναι γεγονότα για κάποιες περιπτώσεις βαφσανισμών ε, στις φυλακές στη Γεωργία. Υπήρχε φωτογραφικό υλικό, το οποίο δημοσιεύθηκε κάποιες ημέρες ε, πριν από τις εκλογές. Και αν θυμάμαι καλά, στο ψήφισμά μας τον περασμένο Νοέμβριο είχαμε ζητήσει από την κυβέρνηση Σεκασβίλη τότε να διερευνήσει το δέμα και να ε, φροντίσει να βελτιωθεί η κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα της Γεωργίας. Ε, με τους πολιτικούς που συναντήσατε και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών συζητήσατε το θέμα. Θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει κάτι στο μέλλον για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. like to ask a colleague. Θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους παρατηρητές αν παρακολούθησαν την κατάσταση αν ήταν και παρόντες, αμέσως μετά την ε, ψηφοφορία και την καταμέτρηση των ψήφων. Σε 11 περιφέρειες, οι εκλογικές επιτροπές φάνηκε ότι ήταν ε, ε, σε κατάσταση ομοιρίας από ε, ομάδες ε, υποστηριχτών του Ιβανιτσβίλη και ε, φαίνεται ότι εκεί το κόμμα το οποίο κέρδισε τις εκλογές ε, δεν έπαιρνε την πλειοψηφία. Υπήρχαν απειλές, θεωρείται ότι κατάφεραν να αλλάξουν τον αριθμό των ψήφων για τους νικητές ή όχι. Και πώς είναι αυτό, πώς δίνει μια εικόνα της δημοκρατίας τα συγκεκριμένα περιστατικά. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji kolegové za Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για όλα τα ερωτήματα τα οποία μου απευθύνατε σχετικά με το γεγονός ότι ένα μέρος της αντιπροσωπείας έκανε χωριστή συνέντευξη τύπου δεν μπορώ να εκφραστώ. Εγώ είχα διαβουλευτεί με όλους τους αντιπροέδρους και όλους τους συναδέλφους και άρα η δικιά μας είναι η επίσημη συνέντευξη τύπου της αντιπροσωπείας όσον αφορά την χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας που ρώτησαν ο κύριος Βαζάιρους Βόλτση και η κυρία Λούνατσεκ ήταν ένα θέμα που συζητήσαμε με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, η Γεωργία έχει πολύ αυστηρή νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και το ελέγξαμε. Και σε 70 περιπτώσεις είχαμε παράπονα τα οποία αντιμετωπίστηκαν και επευλήθησαν σοβαρότατες χρηματικές ποινές, πρόστιμα δηλαδή, ε, για αυτό το γεγονός. Και ε, το, η πλειοψηφία αυτών των παραπώνων ήταν ενάντια, εναντίον του νικητή των εκλογών. Ε, δεν σημαίνει όμως ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμβάλει με τον ίδιο τρόπο σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία όπου υπήρχε μεγάλη πόλωση ε, για να υπάρχει μια πιο ενιαία αντιμετώπιση στο μέλλον θέλω να σχολιάσω ότι η Γεωργία έχει ψηφίσει ένα πολύ καλό εκλογικό νόμο ο οποίος έγινε σεβαστός και όπου οι προϋποθέσεις είναι σαφέστατες. Υπήρξε όντως πολύ μεγάλη πόλωση, υπήρχε ανταγωνιστικότητα, οι άνθρωποι είναι ε, πολύ εκδηλωτικοί ε, και ε, βεβαίως για ένα τόσο σοβαρό θέμα για τη χώρα τους αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχουν εξάρσεις και ε, μπόρεσα να μιλήσω με τον ε, εκπρόσωπο του, του Κοινοβουλίου της Γεωργίας και περιμένω να δω πώς θα κινηθεί το άλλο ίμιση. Επιπλέον θα δούμε πώς θα κινηθούν οι άλλοι συνάδελφοι και θα κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατόν κατά τρόπον οι άλλοι συνάδελφοι να μπορέσουν να κινηθούν στα πλαίσια του Euronest και της συνεργασίας όσον αφορά τις κακομεταχειρήσεις στις φυλακές ε, στις 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 18 μέρες πρώτων εκλογών, ε, υπήρξε μία δημοσίευση στις εφημερίδες σχετικά με αυτό το θέμα που τάραξε τους πάντες ε, και όλοι είχαν ε, πολύ ταραχθεί δύο υπουργοί παρατήθηκαν πολλοί φυλακίστηκαν και οπωσδήποτε αυτό το ο σκάνδαλο επηρέασε πάρα πολύ την έκβαση των εκλογών και πιστεύω ότι η δημόσια γνώμη στη Γεωργία και η πολιτική ε, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τώρα την κατάσταση στις φυλακές και αυτό ε, θα εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει ισχυρότερος έλεγχος και γι' αυτό ε, και εμείς με τους γεωργιανούς ομολόγους μας θα το παρακολουθούμε διότι και αυτοί έχουν συμφέρον τα πράγματα να προχωρήσουν. Κύριε Λαντσμπέργκης ε, ε, ε που όσον αφορά την ε, κατάσταση ε, πρώτων εκλογών ε, υπήρχαν, υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός δύο ώρες πριν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων οι νέοι ήδη γιόρταζαν στους δρόμους νέοι και γέροι με t-shirt του Γεωργιανού Ονείρου ορισμένοι μοίραζαν μπλε σημαίες που είναι ε, το σήμα του κόμματος του Γεωργιανού Ονείρου και είδα πάρα πολλούς πολίτες οι οποίοι ε, γιόρταζαν μετά τις εκλογές. Δεν ε, προσπάθησε κανείς να μας ε, τρομάξει και όλη την ημέρα υπήρχαν παρατηρητές από το κόμμα του Γεωργιανού ονείρου που παρακολουθούσαν και εξασφάλισαν να μην υπάρξει πίεση σε κανέναν ε, επίσης ε, η καταμέτρηση των ψήφων έγινε και κλεισμένων των χωρών χωρίς πιέσεις και ε, υπήρχε ε, ε, ε, υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις από αρμόδιους οργανισμούς και τις οποίες παρακολουθούμε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο για την έκθεση και για την εργασία την οποία έκανε με τους συναδέλφους και τώρα ερχόμαστε στο 17 θέμα της ημερησίας διατάσεως, εργαστήρι σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία εν ώψη των βουλευτικών εκλογών του 2012 και την προετοιμασία των εν λόγω εκλογών. Υπάρχει ένα χωριστό πρόγραμμα και παρακαλώ τον συνάδελφο Κόβαλ να έρθει εδώ. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών και μετά θα συνεχίσουμε.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 herzlich καλωσορίζω σε αυτή τη συνεδρίαση την οποία θα διεξάγουμε από κοινού με τον συνάδελφο Κόβαλ που είναι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας και ε, της ε, Επιτροπής ε, και την αρχή της εβδομάδος με τον κύριο Γκάλερ ε, έκαναν ένα προκαταρτικό ε, ταξίδι στο Κίεβο εάν ε, με έχουν ενημερώσει σωστά. θέλω λοιπόν να τους να τους ενημερώσω κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν να λάβουν το λόγο και οι δύο έρχονται από την Μεγάλη Βρετανία. Πιστεύω ότι από εκεί έχει κανείς την καλύτερη και πιο σαφή εικόνα της κατάστασης. Έχουμε την κυρία Βόλτσουκ από την ε, ε, Birmingham University και η κυρία Μπίρτς από την Essex University. Οπότε έτσι θα μας δώσουν πολύ καλές ε, πληροφορίες και θα μας πούν για τις τελευταίες ε, εξελίξεις στην Ουκρανία και η κυρία Μπέρς για την ε, προετοιμασία για τις εκλογές. Θα έλεγα να ε, ε, κάνει μία εισαγωγή ο κύριος ε, Κόβατς, μετά οι συγητές, μετά θα μιλήσει ο κύριος Γκάλαρ και μετά θα προβούμε στη συζήτηση. Άρα, κύριε Κόβαλ, έχετε το λόγο. Panie Przewodniczący, szczególnie dziękuję za to, że e, znalazł Pan czas na głównym... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε το έτοιμά μου να οργανωθεί η σημερινή ακρόαση και μάλιστα στον τακτικό χρόνο συνεδρίασης της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες ε, που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και ενδιαφέρεται ιδιαίτερο στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα αυτό, καθώς πηγαίνει και μια αντιπροσωπεία ε, του Κοινοβουλίου στη χώρα. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Μπροκ για την ε, ιδέα που είχε να προετοιμαστούμε εγκαίρως μαζί με τον κύριο Γκάλερ. Έχουμε εργαστεί εντατικά για την αντιπροσωπεία προς την Ουκρανία. Έχουμε συναντηθεί με όλες τις ε, πολιτικές παρατάξεις σε συγκεκριμένα πολιτικά επίπεδα και συζητήσαμε για την προετοιμασία των εκλογών. Επίσης μιλήσαμε στους εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ήθελα να τονίσω ότι είχαμε επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για την προετοιμασία των εκλογών με δύο πολύ γνωστές οργανώσεις που παρατηρούν τη διεξαγωγή των εκλογών στην ε, Ουκρανία, την Όπολ, οργάνωση για την παρατήρηση εκλογών και την Επιτροπή για το εκλογικό σώμα της Ουκρανίας. Επίσης έχουμε συναντήσει εκπροσώπους των Ουκρανικών Αρχών, της Αντιπολίτευσης, έχουμε μιλήσει με εκπροσώπους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που διδραματίζει σημαντικό ρόλο στο εκλογικό σύστημα της χώρας. Νομίζω έχουμε συλλέξει ένα σύνολο πληροφοριών διεξοδικό και είμαστε πλήρως έτοιμοι για την βασική αποστολή παρατηρήσεως που θα ξεκινήσει σε δύο εβδομάδες. Το βασικό στοιχείο που θα καθορίσει τη δουλειά μας έχει να κάνει με το πολιτικό τοπίο στην Ουκρανία που βεβαίως θα επηρεάσει τις εκλογές εφόσον κάποιοι από τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να πάρουν μέρος στον εκλογικό αγώνα γιατί αυτή τη στιγμή είναι φυλακισμένοι. Παρατηρήσουμε λοιπόν τις εκλογές για να δούμε κατά πόσο εφαρμόζεται σωστά ο εκλογικός νόμος. Ο νέος ε, νόμος για το, ο νέος εκλογικός νόμος εγκρίθηκε όχι τόσο πρόσφατα. Συνήθως αυτό δεν συνέβαινε στη χώρα, καθώς οι εκλογικοί νόμοι πέρναγαν αμέσως πριν τις εκλογές. Επίσης εδώ πρέπει να πούμε ότι ένα από τα πλεονεκτήματα του νέου εκλογικού νόμου είναι ότι συμφώνησαν και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Τώρα, Κάτι άλλο που συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι περισσότεροι από τους κεφαλείς της ε, αντιπολίτευσης συμφώνησαν με την ε, εφαρμογή του νέου εκλογικού κώδικα και υπάρχουν κάποιες αδυναμίες ε, ως προς αυτή την πτυχή. Εδώ θα πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά τα στοιχεία αυτά που μας προβληματίζουν. Τι εννοώ. το τι θα γίνει με τις ε, περιφέρειες, τις εκλογικές περιφέρειες όπου θα ισχύει η πλειοψηφία. Εκεί υπάρχουν πολλά σχόλια, διότι λέγεται ότι αυτό το τμήμα των εκλογών ε, θα προκαλέσει κάποια επεισόδια. Επίσης, με τις εφορευτικές επιτροπές εδώ υπάρχει ένα, συστηματικό, ένα συστημικό μάλλον σφάλμα σε επίπεδο περιφερειών, διότι είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο για τις ε, για τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να παρατηρήσουν τις εκλογές. Ε, φαίνεται να είναι ένα λάθος νομοθετικό αυτό και το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να το απαλείψουμε. Πώς θα μπορέσουμε να μετριάσουμε τις συνεπειές του πριν τις εκλογές. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα από κοινού με τον πρόεδρο Γκάλερ ότι και πάλι με την αντιπροσωπεία των παρατηρητών ακριβώς πριν τις εκλογές θα συναντηθούμε με τους εκπροσώπους των πολιτικών παρατάξεων και Ίσως η συνάντηση να μην έχει τεχνικό περιεχόμενο πλέον, αλλά θα συναντήσουμε και τους υπευθύνου των διαφόρων εκλογικών κέντρων καθώς και μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Σκοπεύουμε λοιπόν να συζητήσουμε τις αμφιβολίες μας σε σχέση με τον εκλογικό κώδικα και να αποστείλουμε και γραπτές ε, ερωτήσεις προς διευκρίνηση. Οπότε όταν συναντηθούμε και με τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής θα δούμε πώς μπορεί ο εκλογικός κώδικας να βελτιωθεί, να διορθωθεί πριν τις εκλογές. Αυτό που επίσης πρέπει να συζητήσουμε πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, αντικατοπτρίζουν την όλη εκλογική περίοδο και ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, διότι αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένη η πρόσβαση για ορισμένους πολιτικούς κύκλους. Επίσης πώς μπορούν να αγοράζουν διαφημιστικό χρόνο. Ο ρόλος μας σήμερα έγινε στο να εντοπίσουμε ποια είναι τα σημεία που θεωρούμε πλέον ενδιαφέροντα. Δεν θα καταλήξουμε σε απορίσματα σήμερα, ούτε σε συμπεράσματα, διότι θα φτάσει η στιγμή που θα έχουμε παρακολουθήσει την εκλογική διαδικασία στην εξέλιξή τη και τότε θα μπορούμε να έχουμε να διεξαγάγουμε σαφέστερα συμπεράσματα. Θα δούμε κατά πόσο αμέσω πριν τι εκλογέ τα μέσα μαζική ενημέρωση μπορέσαν να παράσχουν πλήρη ενημέρωση και να, να επιτρέψουν την ελεύθερη έκφραση. Μιλάω και για ανεξάρτητου τηλεοπτικού σταθμού μεταξύ άλλων. Θα καλύψουμε όλα αυτά τα στοιχεία πληροφορία και μόλι έχουμε επαρκέ υλικό θα φροντίσουμε να καταλήξουμε σε μια μερόληπτη αποτίμηση του τι συνέβη στην ε, Ουκρανία με τη διεξαγωγή των εκλογών. Όλοι οι πολιτικοί κύκλοι και οι παρατάξεις θέλησαν να μα συναντήσουν στην, από την Ουκρανία. Ε, ζητήσαμε από όλου τους να μας στείλουν και γραπτά σχόλια, ώστε να μπορούμε να τα λάβουμε υπόψη στην τεκμηρίωση της αποτιμησής μας για την εκλογική διαδικασία. Θα ήθελα να καλέσω όσους συμμετάσχουν στην αποστολή παρατήρησης να αξιοποιήσουν το χρόνο πριν τις εκλογές ώστε να συλλογιστούν να παρατηρήσουν τους σημαντικότερους τομείς που σχετίζονται με τις εκλογές. Εκεί όπου μπορεί να προκύψουν ε, ενδιαφέροντα επεισόδια, περιστατικά ε, με σκοπό την προετοιμασία των εκλογών. Νομίζω και ο κύριος Γκάλερ και εγώ περάσαμε αρκετό χρόνο στην Ουκρανία, ώστε να μπορούμε να σα πούμε ποιοι είναι οι τομεί που θα πρέπει να είναι τομεί προτεραιότητα και να του παρακολουθήσουμε στενότερα. Η αποτίμησή μα πιστεύω ότι θα είναι αξιόπιστη. Βεβαίω μετά τη διεξαγωγή των εκλογών. Στο πλαίσιο τη Euronest επίση, οι επαφέ που θα έχουμε θα είναι χρήσιμε, πιστεύω και είναι πολύ εκείνοι που ενδιαφέρονται για την Ουκρανία, όχι μόνο όσοι θα συμμετάσχουν στην παρακολούθηση την αποστολή δηλαδή παρατήρηση των εκλογών. Αλλά σήμερα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τι θα πρέπει να παρατηρήσουμε σε σχέση με την προηγούμενη διεξαγωγή των εκλογών το 2010 και τις προεδρικές καθώς και τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Τα πράγματα έχουν αλλάξει εδώ μεταξύ στην Ουκρανία. Θα δούμε κατά πόσον ο εκλογικός νόμος είναι δημοκρατικότερος, κατά πόσον είναι πιο προοδευτικός, ευρύτερος και καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών. Μπορούν οι πολίτες να επιλέξουν ελεύθερα τους εκπροσώπους τους ή το ανάποδο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω ξανά σήμερα τον ε, πρόεδρο Μπροκ που επέτρεψε να διοργανωθεί αυτή η συζήτηση και να ευχαριστήσω και τους προγνώμονες που είναι μαζί μας. Δεν θα είναι τελευταία μας συνάντηση και οι απόψεις θα προλυάνουν το έδαφος για να ερμηνεύσουμε σωστά την πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία ως αποστολή παρατήρησης. Θα παρακολουθήσουμε στενά τις εκλογές, αλλά όχι μόνον. Θα ασχοληθούμε και με το ευρύτερο πολιτικό τοπίο στη χώρα, με την αποστολή Κροσνεύσκη και Κόξ. Ποτέ στην ιστορία μας. Δεν δείξαμε τόσο ενδιαφέρον ε, για την Ουκρανία και τη σχέση με τη χώρα αυτή. Η αποστολή λοιπόν ε, θα βασιστεί στην Επιτροπή για την Κοινοβουλευτική Συνεργασία, στη σημερινή συνάντηση, στην Αποστολή Κρυφέσκη Κόξ και σε άλλες πρωτοβουλίες των πολιτών. Σας ευχαριστώ και να δώσω πάλι το λόγο στον Πρόεδρο. Θα ξεκινήσουμε τώρα με την κυρία Κατερίνα Βόλτσικ. Thank you very much for the... Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Φαίνεται ότι με περιβάλλει τεχνολογία και ζητώ συγγνώμη για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσω εγώ εκ των προτέρων. Νομίζω ότι βρίσκομαι στην καλύτερη ε, θέση για να συζητήσω το θέμα της Ουκρανίας. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη για την Ουκρανία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλαβαίνει απόλυτα ε, την Ουκρανία. Ε, είναι, υπερβαίνει και αρκετά ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα. Επομένως δεν πηγαίνω σε κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το θέμα. Θα προσπαθήσω παρόλα αυτά να σας παρουσιάσω μια ευρύτερη εικόνα, να σας ε, δω πώς έχει το ιστορικό και κάποιες πιθανές ε, συνέπειες λόγω των όσων συμβαίνουν, ε, έχουν συμβεί στο παρελθόν. Έχουμε εδώ ένα χάρτη της Ουκρανίας και θα ξεκινήσω εν συντομία με τις πολιτικές εξελίξεις. Ε, δεν θα σας ε, καθυστερήσω. Ε, θα σας πω απλώς ε, τι έχει συμβεί από τον Ιανουάριο του 2010 και τις προηγούμενες εκλογές. Τι είδαμε, ότι έχουμε μια συνταγματική αποκατάσταση εντός εγωγικών του ρόλου του Προέδρου. Ε, και στη μετά σε βιωτική εποχή ε, αυτό αποκαλείται η συνιστόσα της εξουσίας ε, από την Προεδρία. Και αυτό φυσικά πηγαίνει από τον Πρόεδρο σε περιφερειακό επίπεδο και έχει σχέση και με το Σύνταγμα ε, το οποίο αναβιώθηκε το 2010 από το 1996 που είχαμε αρχικώς αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι μειωμένη πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, έχουμε ε, κάλυψη προεκλογικής ε, εκστρατείας από τις, ε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μειωμένη πολυφωνία. Γιατί συμβαίνει αυτό. Ε, υπάρχουν κάποιες ε, ε, πιέσεις για τη χρήση των διοικητικών πόρων όπως αποκαλούνται. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες να ποινικοποιηθεί η δυσφήμιση από τους δημοσιογράφους, αλλά υπάρχει και μια κρισία. Ε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τις εκλογές, τις καλύπτουν κατά τρόπον ε, ώστε, όπως θεωρούν αυτοί, ε, να γίνουν αποδεκτές ευνοϊκά. Και αυτό φυσικά είναι αρνητικό στοιχείο και, ε, και για τις προσδοκίες των πολιτικών παραγόντων στην Ουκρανία. Είναι ουσιαστικά μια αυτοεπληρούμενη προφητεία. Πέραν αυτού βέβαια δεν είναι τα πάντα έτσι. Υπήρξαν κάποια παραδείγματα και πρέπει να τα τονίσουμε. Έγινε μια πρόσφατη απόπειρα να περάσει ένας νόμος για τη δυσφήμιση από κάποια μέλη της, ε, του Κοινοβουλίου από το Κόμμα των Περιφερειών και υπήρχαν και αντίστοιχες απαντήσεις από τους δημοσιογράφους και αυτό δείχνει ότι ε, αρχίζει να προωθείται η κοινωνία των πολιτών και το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν πλέον να διαδηλώσουν ε, ε, είχε ως αποτέλεσμα αυτό το σχέδιο νόμου προς το παρόν να μπει ε, στο περιθώριο. Αν περάσουμε λοιπόν από το πολιτικό πλαίσιο τώρα στην οικονομική απόδοση, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον υπάρχει συγκεκριμένη οικονομική απόδοση που να είναι σημαντική για τις επόμενες εκλογές. Αυτό που είναι σημαντικό για τον πρόεδρο Γιαννουκόβιτς είναι ε, ότι όταν ε, ανέλαβε την εξουσία το 2010 είχε εντολή ουσιαστικά να βελτιώσει την ε, οικονομία. Αυτό επειδή υπήρχαν προβλήματα μετά από την οικονομική κρίση του 2008 και η Ουκρανία ήταν μία από τις χώρες που χτυπήθηκαν περισσότερο. Ε, η Αρμενία χτυπήθηκε με 14%. Είδαμε μια κάποια ανάκαμψη, αλλά όχι όσο ήταν αναμενόμενη και όχι όσο περίμενε και το εκλογικό σώμα. Η εντολή ουσιαστικά που δόθηκε στον πρόεδρο Γιανοκόβιτς και στον κόμμα των περιφερειών δεν εκπληρώθηκε για αρκετούς λόγους, ε, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολύ μεγάλες προσδοκίες από πλευράς ε, κοινού. Βέβαια, κανένα πολιτικό κόμμα στην ε, Ουκρανία δεν έχει καλό ιστορικό για τη διαχείριση των οικονομικών παρά τις προσδοκίες των Ουκρανών πολιτών. Δεν υπάρχουν λοιπόν κόμματα που να έχουν ε, ε, μεγαλύτερη αξιοπιστία, είτε γιατί όταν ήταν ε, στην εξουσία δεν έγιναν οι κατάλληλε οικονομικέ μεταρρυθμίσει, ή γιατί κάποιοι όπω το Ουντάρ δεν έχουν δοκιμαστεί στην κυβέρνηση. Να δούμε λίγο τώρα το κόμμα των περιφερειών, το κυβερνών κόμμα. Παρά τα όσα έχουν ακουστεί για το κόμμα αυτό και τις αρχές, είναι σαφές ότι και ο πρόεδρος Γιαννοκόβιτς και το κόμμα των περιφερειών προσπαθούν να εξασφαλίσουν διεθνή νομιμοποίηση. Και φυσικά ε, θέλουν να επιβεβαιώσουν ότι αυτές οι εκλογές ε, ε, θα γίνουν με βάση τις ε, ε, πάγιες διεθνείς πρακτικές. Και γιατί προσπαθούν να εξασφαλίσουν αυτή τη διεθνή νομιμοποίηση. Γιατί το κόμμα των περιφερειών θέλει να εδραιώσει την εξουσία του εντός της Ουκρανίας και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ως φαινόμενο, διότι πέραν της Προεδρίας αυτό που απαιτείται είναι να υπάρχει και κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες ενδιαφέρουσε εξελίξεις εντός του κόμματος. Ε, έχει σημειωθεί ότι ε, ανεβαίνει η λεγόμενη οικογένεια στην Ουκρανία. Αυτή είναι μια πρόσφατη έννοια. Η Ουκρανία δεν είχε ε, περιστατικά οικογενειακής πολιτικής όπως το Αζερβαϊτσάν για παράδειγμα. Ε, είναι ένα καινοφανές στοιχείο στην Ουκρανία και δεν μπορούμε ακόμα να το ερμηνεύσουμε παρκώς. Αλλά παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κατηγορίες για την οικογένεια του Προέδρου Γιαννικόβιτς, ε, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλη συνοχή στο κόμμα των περιφερειών, ε, ε, ιδίω και σε σύγκριση με την αντιπολίτευση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα πολιτικά κόμματα της Ουκρανίας. Και κάτι ακόμα το οποίο διαπιστώσαμε, παρά το γεγονός ότι δεν είναι καλή οικονομική απόδοση της Ουκρανίας, είναι ότι το κόμμα των περιφερειών έκανε μια πολύ αποτελεσματική εκλογική, προεκλογική εκστρατεία και θεωρείται από τις καλύτερες μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και σύμφωνα με κάποιο δημοψήφιο ψήφισμα ε, ε, που έγινε μεταξύ 50 Ουκρανών εμπειρογνωμόνων ε, θεωρείται από τις καλύτερες. Επίσης, ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι το γλωσσικό ζήτημα και η εξέταση της γεωγραφικής πόλωσης στην Ουκρανία. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Θα σας δείξω και κάποιους χάρτες που δείχνουν ότι οι προτιμήσεις ψήφου ε, σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις εθνικές και γλωσσικές ε, διαιρέσεις. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις τωρινές εκλογές, αλλά είναι μια μακροπρόθεσμη τάση στην Ουκρανία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ο νόμος για τη γλώσσα ο οποίος αποτέλεσε το ένευσμα για διαδηλώσεις και βία στην Ουκρανία είναι τμήμα της εκστρατείας ε, θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ε, για να εδραιώσει τη θέση του κόμματος των ε, περιφερειών. Να ρίξουμε λοιπόν μια γρήγορη μακριά στην εθνοτική σύνθεση της Ουκρανίας σύμφωνα με μια την πρόσφατη απογραφή του 2001. Από ό,τι βλέπουμε οι Ρώσοι στην Ουκρανία είναι στα νότια και ανατολικά τμήματα και αυτό σχετίζεται και με τον τρόπο με τον οποίο μιλείται η γλώσσα. Η διέρεση είναι σχεδόν πανομοιότυπη, δηλαδή το βλέπετε και στο χάρτη, έχουμε τις εκτιμήσεις, δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε σε λεπτομέρειες ε, τα αριθμητικά στοιχεία, θα δείτε απλώς τα χρώματα στο χάρτη η ρωσική γλώσσα κυριαργεί στα νότια και ανατολικά τμήματα της Ουκρανίας και ο πρόσφατος νόμος για τη γλώσσα ουσιαστικά αναγνωρίζει επισήμως ε, τη ρωσική ως ε, επίσημη γλώσσα. Τώρα, υπήρχαν οι, λεγόμενες, οι αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές ε, στην Ουκρανία και εδώ βλέπετε ότι τα χρώματα στο χάρτη συμπίπτουν και πάλι με ε, τον τρόπο με τον οποίο κατανεμήθηκαν οι ψήφοι στο, ε, στα διάφορα τμήματα της χώρας. Το δυτικό τμήμα ήταν βασικό για την ήχη του, ε, της Γιουσένκο και ο κύριος Γιανουκόβιτς κέρδισε στα νότια και ανατολικά της χώρας. Όλα αυτά ήταν προβλέψιμα. Εδώ ε, έχουμε τα ίδια σχεδόν αποτελέσματα και στις προεδρικές εκλογές ε, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά υποπροϊόντα της ε, πορτοκαλία Επανάστασης. Υπάρχει μια σαφής κατανομή αναπεριφέρειας ουσιαστικά στην Ουκρανία. Αν βέβαια εξετάσουμε τα πράγματα λίγο βαθύτερα, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και εδώ έχουμε τα αποτελέσματα των τελευταίων κοινοβουλευτικών εκλογών στην Ουκρανία, που δείχνουν τα αποτελέσματα των ε, κομμάτων που βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις. Το μπλε είναι το κόμμα των περιφερειών και μετά το μοφ, ή μάλλον κόκκινο όπως φαίνεται εδώ στην οθόνη, είναι το ε, Fatherland, ε, τότε αποκαλούνταν Μπιούκ και είναι το κόμμα της Γιούλια Τιμοσέγκου. Αυτό δείχνει ότι είναι πολύ ισχυρές αλλά διαφορετικές προτιμήσεις, αλλά εάν εξετάσουμε λίγο βαθύτερα τα πράγματα, βλέπετε ένα, δέσκολο, ένα χάρτη για ε, όσους βρέθηκαν στη δεύτερη θέση και εδώ βλέπουμε ότι ο συνασπισμός της Γιούλια Τιμοσέγκου ήρθε δεύτερη ε, σε αρκετές ε, περιφέρειες στην ε, Νότια και Ανατολική Ουκρανία. Υπάρχει λοιπόν πεδίο για το συνασπισμό της Γιούλιαν Τιμοσέγκο και θα μπορούσε ίσως να γίνει εθνικό κόμμα το οποίο να έχει επιρροή σε όλη την Ουκρανία. Τώρα όμως έχουν ξαναπάει τα πάντα ε, στο μηδέν και δεν ξέρουμε πώς θα καταναμηθούν ε, τα κόμματα. Υπάρχει ένα ε, νέο κόμμα όπως για παράδειγμα το Ουντάρ ή και το Fatherland. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να διατηρήσουν την ίδια ισχυρή παρουσία στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας ή αν θα επανέλθουμε στην ισχυρή πόλωση μεταξύ των δύο πλευρών της Ουκρανίας. Ο γλωσσικός νόμος φαίνεται ότι ο στόχο είχε να εδραιώσει την επιρροή και να διατηρήσει την εξουσία του κόμματο ε, των περιφερειών στη νότια και ανατολική ε, Ουκρανία και να αποκλείσει ουσιαστικά άλλα κόμματα. Τώρα, να ρίξουμε μια πιο ε, στενή ματιά στις ε, εκλογές αυτές καθ' αυτές. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες στην Ουκρανία, και αυτό επιβεβαιώνεται και από στοιχεία δημοσκοπήσεων, τέσσερα κόμματα αναμένεται να υπερβαίνουν το όριο του 5% στις ε, λίστες των εκλογών. Ε, βάσει του εκλογικού νόμου αποκλείονται οι συνασπισμοί κομμάτων και επομένω τώρα έχουμε τέσσερα κόμματα. Ουσιαστικά ο εκλογικό ε, νόμος βοήθησε την αλλαγή του συστήματος των κομμάτων. Έχουμε το κόμμα των περιφερειών, το Fatherland, το Ουντάρ και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπάρχουν αρκετά, αρκετά, αρκετές δημοσκοπήσεις, ε, μία από το Σεπτέμβριο του 2012, με κάποιο περιθώριο σφάλματος φυσικά, εντός του περιθωρίου σφάλματος, φαίνεται ότι το κόμμα των περιφερειών βρίσκεται μπροστά, ε, το Fatherland και το Ουντάρ ε, ακολουθούν. Ε, και κάποιοι θεωρούν ότι ανεβαίνουν κιόλα και το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει κάνει μια πολύ καλή επάνωδο, η οποία θα μπορούσε να σχολιαστεί κι αυτή ε, ίσως λίγο αργότερα. Να δούμε τώρα την αντιπολίτευση. Εδώ ουσιαστικά έχουμε δύο κόμματα, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη αντιπολίτευση στο κόμμα των περιφερειών και ε, γιατί ε, ουσιαστικά η ισχύ τη είναι στα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας. Τώρα, το Fatherland όμως ε, και το Ουντάρ είναι πιο ισχυρά κόμματα και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ε, το κόμμα Fatherland επειδή κάποια βασικά πολιτικά προ, ε, πρόσωπα πέρασαν δίκη και γιατί ο νέος πρόεδρος του κόμματος είπε ότι δεν έχω το χάρισμα Τη Γιούλια Τιμοσέγκο και φυσικά αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις εκλογές. Το γεγονός βέβαια ότι τα βασικά πρόσωπα του κόμματος ε, αμφισβητούνται είναι σημαντικό για, την, ε, για το κόμμα αυτό η εκστρατεία τους δεν θεωρώθηκε και πάρα πολύ αποτελεσματική από τους Ουκρανούς εμπειρογνώμονες. Ο, ο νέος, ε, ο νέος ερχόμενος είναι το κόμμα Ουντάρ, ε, ξεκίνησε από μια ανεξάρτητη προεκλογική εκστρατεία, αρνήθηκε να ενταχθεί στο Fatherland παρά τις πάρα πολλές εκκλήσεις και υπάρχουν αρκετοί ανεξάρτητοι ε, υποψήφοι στις ε, βασικές ε, ε, περιφέρειες όπου υπάρχει πλειοψηφία. Και από, κάποια, ε, από κάποιες δημοσιοσκοπήσεις φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει την Γιούλια Τιμοσέγκο στην, ε, στην κούρσα για τις εκλογές. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και οι εκλογές του 2015 για την εκλογή Προέδρου, που είναι το βασικό στοιχείο και οι παρούσες εκλογές φαίνεται ουσιαστικά να προλύνουν το έδαφος για τις επόμενες εκλογές το, γενικό, το γεγονός ότι ο Κίτσκο φαίνεται να είναι ε, ανερχόμενος υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές μπορεί να πιέσει και το κόμμα του να κάνει ένα συνασπισμό ή μια συμμαχία με το Fatherland ε, αυτή στιγμή συνταχθούν στο κοινοβούλιο όπως αναμένεται αυτή τη στιγμή. Κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό είναι ότι η αντιπολίτευση αντιλαμβάνεται με πολύ πολλωμένο τρόπο την πολιτική κατάσταση και υπάρχει πολύ μεγάλη ε, έλλειψη εμπιστοσύνης ε, για τις αρχές ε, από τους εκπροσώπους των δύο κομμάτων. Υπάρχει αυτό λοιπόν το λεγόμενο vertical της εξουσίας, το οποίο έχει επηρεάσει τη στάση που τηρούν αυτά τα κόμματα και το πώς διεξάγουν από εκεί και πέρα την προεκλογική τους εκστρατεία. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Εδώ έχουμε μία, ε, ένα διάγραμμα από μία δημοσκόπηση. Δεν θεωρώ βέβαια ότι αυτό που βλέπετε θα είναι αποφασιστική σημασία για το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπίτς τώρα έχει το λόγο. Α, νόμιζα ότι τελειώσατε. Ε, καταφέρατε να με μπερδέψετε. Παρακαλώ, συνεχίστε. Δύο λεπτά, εντάξει. Για τις εκλογές, λοιπόν. Ε, Εξαιτία της δυσπιστίας και παρόλο που η αντιπολίτευση έχει συμφωνήσει με το νέο εκλογικό σύστημα οι εκλογές γίνονται σε πολύ ε, μεγάλη ένταση, ε, πολιτική ένταση. Και εδώ υπάρχουν λεπτομέρειες του εκλογικού νόμου που αμφισβητούνται από όλου. Αυτό είναι κλασικό στην Ουκρανία. Ε, πρώτα απ' όλα συμφωνούν στο νόμο γενικώ και μετά διαπιστώνουν τις ασυνεπείς τι λεπτομέρειε. Οπότε αυτό μπορεί να δώσει και λαβή για τις ε, μετεκλογικές διαφορές που θα προκύψουν τα παράπονα ή τις προσφυγές. Ποιε είναι οι πιθανότητε τώρα, και αυτό που προσπαθώ εγώ να κάνω είναι να σα παρουσιάσω μια εικόνα που είναι αρκετά περίπλοκη στην πραγματικότητα. Διότι οι δημοσκοπήσεις ω τώρα δεν είναι αντιπροσωπευτικέ. Δεν μα λένε τι αποτέλεσμα θα μπορούσαμε να έχουμε κατάλογοι, οι εκλογικοί κατάλογοι έχουν, οι εκλογικές λίστες έχουν ε, προσελκύσει την ε, προσοχή, παρατηρούνται με προσοχή από τα μέσα μαζικής ενημέρωση και πιστεύετε ότι η αντιπολίτευση θα τα πάει καλύτερα από ότι το κόμμα των περιφερειών. Ωστόσο, το μέλλον των εκλογών θα καθοριστεί από τις μονεδρικές περιφέρειες. Υπάρχουν πολλοί υποψήφοι, πάρα πολλοί, αυτό βεβαίως και μπερδεύει ακόμη περισσότερο τους ε, ψηφοφόρους. Οι περισσότεροι έχουν διοριστεί από τα κόμματα, όμως το 45% ένας μεγάλος αριθμός είναι ανεξάρτητοι. Ε, αναμένεται επίσης μεταξύ των εμπειρογνωμόνων τα κόμματα της αντοπολίτευσης να τα πάνε χειρότερα στις μονεδρικές περιφέρειες. Και ακριβώς επειδή αυτό το σύστημα ισχύει κατά αυτόν τον τρόπο, αυτό θα καθορίσει και το αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μεγάλη αστάθεια λόγω και των προηγούμενων εμπειριών μας με τις κοινοβουλευτικέ εκλογές. Αυτό που πιθανώς να συμβεί είναι να υπάρξουν μετατοπίσεις μετά τις εκλογές, δηλαδή διάφορα κόμματα να προσελκύσουν ανεξάρτητους βουλευτές. Αυτό συνέβη και στο παρελθόν και αυτό που που συμβαίνει είναι ότι ακριβώ λόγω των δημοσκοπήσεων είναι αδύνατο να προβλέψουμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά ακόμη και έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την ε, ισορροπία του ποιο έχει την εξουσία και πάλι τον έλεγχο έχει ο πρόεδρο. Το σύνταγμα είναι σαφέ. Η ε, Ουκρανία έχει ένα ημιπροεδρικό σύστημα όπου επιτρέπεται στον πρόεδρο να διορίζει τον, να ονομάζει τον πρωθυπουργό, να τον προτείνει. Δηλαδή οι εκλογές είναι σημαντικές, αλλά είναι δύσκολο να δημιουργηθούν ίσοι κανόνες παιχνιδιού και να προβλεφθεί το τι ακριβώς θα γίνει στις προεδρικές εκλογές του 2015. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. E, και τώρα η κυρία Μπίρτς. Um, σας ευχαριστώ. Μετά τη συζήτηση για το γενικό πολιτικό τοπίο στην Ουκρανία που σας παρουσίασε η κυρία Βόλτσουκ, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον εκλογικό νόμο με τη σειρά μου και μερικά από τα βασικά στοιχεία που έχουν προκαλέσει ανησυχίες σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, τα διεθνή πρότυπα, τις βαλτιστές πρακτικές και τα εκλογικά πρότυπα καθώς και τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ουκρανίας. Πολύ σύντομα να ξεκινήσω παρουσιάζοντας το ιστορικό για να δούμε την έννοια της εκλογικής ακεραιότητας όπως ονομάζεται. Υπάρχουν διαφορετικέ δεσμεύσει που έχει αναλάβει κάθε δημοκρατική χώρα βάσει του διεθνούς δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να στρεβλωθούν τα εκλογικά αποτελέσματα με τρεις ε, διαφορετικούς τρόπους, ενδεχομένως. Αυτό, εάν ε, παραβιαστεί ο εκλογικός νόμος ή στρεβλωθεί έτσι ώστε να αντίκειται στο διεθνές δίκαιο ή εφόσον χειραγωγηθεί η εκλογική εκστρατεία και παραβιάζει τα διεθνή πρότυπα και βεβαίως μπορεί να υπάρξει και στρέμλωση εφόσον ε, η διαδικασία της εκλογικής αναμέτρησης υπονομευθεί. Και αντίκειται και πάλι στα διεθνή πρότυπα. Πρέπει εδώ να ε, τονίσουμε ότι εάν οποιαδήποτε από αυτά τα τρία στοιχεία είναι αρκετά σοβαρό, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι αμφισβητούμενο το εκλογικό αποτέλεσμα. Η εκλογική ακεραιότητα, νομιμότητα μάλλον και η αξιοπιστία δεν απλά ζητήματα. Δεν είναι θέμα αμφισβήτησης απλώς ή αν είναι ελεύθερε οι εκλογές. Τώρα να δούμε συγκεκριμένα την Ουκρανία. Μια ανασκόπηση του εκλογικού συστήματο ε, και το τι έχει γίνει με τι βουλευτικέ εκλογέ ω τώρα στην Ουκρανία. Από το 1990 στο 1994 είχε το σοβιετικό ε, σύστημα η Ουκρανία με το μονοεδρικό σύστημα περιφερειών με απόλυτη πλειοψηφία. Το 1998 με 2002 πέρασε σε ένα παράλληλο μεικτό σύστημα. Οι μισέ έδρε κατανείμονταν με αναλογική κεντρικέ εκλογικέ λίστες, είναι οι υπόλοιπε με τι μονοεδρικέ. και από το 2006 έω το 2010 ε, και πάλι υπήρξε αναλογική αντιπροσώπευση με ένα όριο 3%. Το 2012 υπήρξε μια επιστροφή, όπως είπε και η δόκτωρ Βόλτσεκ, στο ε, μεικτό παράλληλο σύστημα που είχε η Ουκρανία από το 1998 στο 2002. Οι 140 έδρες ε, πληρούνται από τους αναλογικούς ε, εκλογικούς λίστε. λίστες τι αναλογικέ εκλογικέ λίστε, το 50% από τι μονοεδρικέ και υπάρχει και ένα όριο 5%. Όμω δεν υπάρχουν συνασπισμοί κομματικοί που να μπορούν να λάβουν μέρο στι εκλογέ, ενώ ε, οι υποψήφοι δεν μπορούν να λάβουν μέρο και στι μονοεδρικέ αλλά και στι ε, αναλογικέ εκλογικέ λίστε. Η επιστροφή στο μεικτό σύστημα θεωρήθηκε στι εκλογέ τοπικέ αυτο... το 2010 ως μια αρνητική τροπή. Και δημιουργήθηκαν αρκετές αμφιβολίες ε, σε διεθνές επίπεδο για την διεξαγωγή των εκλογών. Κυρίως λόγω της ε, πρόσβασης, ε, δηλαδή κανόνες που επιτρέπουν στους υποψηφίους να φτάσουν ως την πρότασή τους, την υποψηφιότητά τους, το πώς φτάνουν ως την κάλπη. Αμφισβητήθηκε λοιπόν το εκλογικό σύστημα ιδίω και για τους κομματικού συνασπισμού. Υπάρχουν λοιπόν ανησυχίε για το τι θα συμβεί με τι κοινοβουλευτικέ εκλογέ του 2012. Άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κοινοβουλευτικέ εκλογέ στι 28 του μήνα. Πρώτα απ' όλα το εκλογικό σύστημα. Η Επιτροπή της Βενετίας και ο ΑΣΕ ε, εξέδωσαν μια έκθεση για τον εκλογικό νόμο πέρσι και σχολίασαν ζητήματα που ακόμη δεν έχουν επιληθεί. Πρώτα απ' όλα την απαγόρευση για τους κομματικούς συνασπισμούς. Είναι ασαφές πώς αιτιολογείται μια τέτοια απαγόρευση. Ιδίως από δημοκρατικής άποψης. Έπειτα η έλλειψη σαφών κριτηρίων για, τα, για τον ορισμό των περιφερειών και τα σύνορά τους η διακριτική ευχέρεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για το πώς ε, θα οριστούν οι περιφέρειες. Δεν υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμέ και έγιναν κάποιες μελέτες για τα όρια που είχαν ήδη επιλεγεί για τις μονεδρικές περιφέρειες, αλλά αυτά δεν είναι ακόμη τελεσίδικα. Πολλέ φορέ ο καθορισμό των συνόρων γίνεται για να ευνοηθούν ε, κάποια κόμματα. Ένα άλλο ενδεχόμενο πρόβλημα που σχετίζεται με την επιστροφή των μονοεδρικών είναι η δυνατότητα στρέβλωσης των ορίων ακριβώς. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα ε, ενιαίο για όλο το έθνος σύστημα αναλογικής αντιπροσώπευσης. Επίσης, για τη χρηματοδότηση των εκλογικών εκστρατιών, οι κανόνες αυτοί έχουν επικριθεί. Δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια. Τα κόμματα μπορούν να λάβουν τα χρήματα από θέλουν, να τα δαπανίσουν όπω θέλουν. Ο δημοσιονομικός κανονισμός είναι πολύ ασαφή. και ο γενικό κανονισμό στην Ουκρανία είναι υπανάπτυκτο ακόμα. Επίσης, η έκθεση της Επιτροπής της Βενετίας αναφέρεται και στα όρια για το δικαίωμα να θέσει κανείς υποψηφιότητα, στους περιορισμούς που επιβάλλονται. Ιδίω εάν κάποιο έχει καταδικαστεί ή βρίσκεται στη φυλακή. Αυτό το ζήτημα προφανώ είναι αμφιλεγόμενο, αλλά βλέπετε εδώ ένα απόσπασμα της ίδιας της έκθεσης που λέει ότι ο περιορισμός ε, στο δικαίωμα ψήφου για γενικές ε, κατηγορίε ομάδων πολιτών, χωρί να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά περιστατικά και χαρακτηριστικά που αφορούν το συγκεκριμένο άτομο, δεν συνάδουν με το διεθνέ δίκαιο. Η ε, άρνηση του δικαιώματο να θέσει κανεί υποψηφιότητα κάποιου που έχει καταδικαστεί ή διαπράξει εγκληματική ενέργεια θα πρέπει να είναι τόσο σοβαρή ώστε η στέρηση του πολιτικού δικαιώματος να είναι του πολιτικου δικαιώματο να ειναι λογικη με το ε, έγκλημα που έχει διαπραχθεί. Όλες αυτές οι ανησυχίες που εντοπίζει, εντοπίζονται σε σχέση με τον εκλογικό νόμο ε, έχουν εκτεληθεί και στην εκλογική εκστρατεία όπως έχει διεξαχθεί ως τώρα. Υπάρχουν λοιπόν ανησυχίες για τις ίδιες εκλογές και την εξαγωγή τους. Πρώτα απ' όλα, πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε αν θα θεωρηθούν νόμιμες και ελεύθερες οι εκλογές εφόσον η κυρία είναι στη φυλακή. Υπάρχουν δύο στοιχεία εδώ. Πρώτα απ' όλα, Όπω η Επιτροπή τη Βενετία και ο ΑΣΕ εντόπισαν, εάν κάποιο είναι φυλακισμένο, προφανώ δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Αυτό ίσω να είναι ευθύ εξ αρχή παραβίαση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Αλλά εφόσον πρόκειται και κοινοβουλευτικέ εκλογέ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είχαν καμία δυνατότητα να συμμετάσχουν στι εκλογέ, το ερώτημα είναι το εξή. Τι σημασία έχει εάν κάποια περιορισμένα, ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές. Για στις 156 έδρες του Κοινοβουλίου δηλαδή. Έπειτα, πώς μπορεί ένα κόμμα να προωθήσει την υποψηφιότητά του εν επικεφαλής του κόμματος δεν ε, μπορούν να διαδραματίσουν το ρόλο που τους αναλογεί η ε, στέρηση ελευθερίας της έκφρασης επηρεάζει εδώ την λειτουργία της αντιπολίτευσης και της πραγματικής ε, εκλογικής εκπροσώπηση σε μια εκλογική εκστρατεία. Αυτό έχει διαφορά από τη στέρηση του δικαιώματο ε, ψήφου. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η δυνατότητα των κομμάτων να κάνουν την εκλογική εκστρατεία που θέλουν. Και αυτό ίσω να είναι και σοβαρότερο από την μεμονωμένη υποψηφιότητα ενός συγκεκριμένου ατόμου. Εδώ δεν μιλάμε για προεδρικέ εκλογέ. Για προεδρικέ εκλογέ ίσω να ήταν σοβαρότερο να στερούνται τα δικαιώματα αυτά από ένα συγκεκριμένο άτομο. Εδώ όμω, εφόσον πρόκειται για κοινοβουλευτικέ εκλογέ, το θέμα είναι κατά πόσο είναι αποτελεσματική η εκλογική εκστρατεία. Και ιδίω εφόσον οι επικεφαλεί ενό κόμματο βρίσκονται στην φυλακή. Έπειτα, η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό το έθεσαν και ο κύριος Κοβάλ και η κυρία Βόλτσοκ. Εδώ φαίνεται να ασκείται ε, εκφοβισμός και παρενόχληση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν υπάρχει πρόσβαση για τα διάφορα κόμματα, το είπε και η κυρία Βόλτσουκ, υπάρχει αυτολογοκρισία και κάτι που έχουν αναφέρει πολλοί που παρατηρούν την εκλογική εκστρατεία στην Ουκρανία λένε ότι υπάρχει πολλής φόβος, φόβο για τα μέσα σαν στην Ουκρανία. Τα μέσα δεν μπορούν να ασκήσουν την ελευθερία έκφραση που θα έπρεπε να διαθέτουν και δεν μπορούν να καλύψουν την εκστρατεία με τρόπο μερόληπτο. Επίση υπάρχει και κάτι ακόμη που ανέφερε η δόκτωρ Βολτσούκ, η χρήση διοικητικών πόρων Οι κρατικές δυνατότητες εδώ είναι σίγουρα υπερβατικές. Δηλαδή υπάρχει κατάχρηση των κρατικών πόρων προκειμένου οι παρτιζάνοι ενός του κρατικού κόμματος, να, του κόμματος του κυβερνώντος να εποφελούνται. Όσοι βλέπουν τι γίνεται με την εκλογική εκστρατεία επιτόπου λένε ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα σε αυτές τις εκλογές. Κάτι άλλο που ο κ. Κοβάλ σχολίασε είναι το τι γίνεται με την εκπροσώπηση στι εφορευτικέ επιτροπέ. Το πώ σχηματίζονται οι εφορευτικέ επιτροπέ. Τα περισσότερα κόμματα τη αντιπολίτευση δεν έχουν καθόλου πρόσβαση. Δεν αντιπροσωπεύονται. Και αυτό βεβαίω εγείρει ανησυχίε. για το πώς τελικά μπορεί να λειτουργήσουν την ημέρα των εκλογών οι εφορευτικές επιτροπές. Η μέρα των εκλογών τώρα, αυτή καθεαυτή. Εκεί μπορεί να προκύψουν άλλα ζητήματα. Μια εξέλιξη, κάτι το καινούργιο στην Ουκρανία σε αυτές τις εκλογές, είναι τοποθέτηση ε, κάμερας, webcam, στους στα διάφορα εκλογικά κέντρα. Το είδαμε αυτό και αλλού στο παρελθόν, στο Αζερβαϊτζάν, στη Γεωργία. Ίσως έτσι να περιοριστεί η νοθεία και να εξασφαλιστεί περισσότερη διαφάνεια ενδεχομένως να πετύχει κάτι το μέτρο αυτό, όμως δεδομένου του κόστους ...124.000 δολάρια ακούστηκε πρόσφατα. Δεδομένου λοιπόν αυτού του κόστους... ...δεν ξέρω κατά πόσο να εξυπηρετούν οι κάμερες αυτές του διαδικτύου εφόσον το πεδίο που καλύπτουν είναι περιορισμένο και μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Βεβαίω θα υπάρχουν πάντοτε περιοχέ και σημεία στο εκλογικό κέντρο που δεν θα καλύπτονται. Δεν μπορεί τα πάντα να τα καλύψει μια κάμερα. Επίση, δεν καλύπτουν όλε τι πτυχέ τη εκλογική διαδικασία. Την καταμέτρηση των ψήφων, την ε, σωστή καταγραφή των ε, ψηφισάντων. Επίσης, τελικά μπορεί οι επιπτώσεις από τη χρήση τους να μην είναι οι αναμενόμενες, ο περιορισμός της νοθεία λόγου χάρη. Υπάρχει όμως και άλλο ζήτημα σχετικά. Οι μελέτες για τη χρήση των ε, συστημάτων αυτών και σε άλλες χώρες στο παρελθόν δείχνουν ότι κάποιοι αποθαρρύνονται, οι πολίτες αποθαρρύνονται από το να πάνε να ψηφίσουν λόγω της χρήσης της κάμερας. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι ο εκλογικός νόμος αποδίδει αμφίσιμες εξουσίες στους παρατηρητές, τους εγχώριους παρατηρητές των εκλογών να εμποδίσουν παράνομες ενέργειες στι διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Αυτό που ορίζεται για τους παρατηρητές είναι ότι σε καμία περίπτωση αυτοί δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στην εκλογική διαδικασία. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο νόμος που επιτρέπει στις ε, εφορευτικές επιτροπές των συγκεκριμένων κέντρων να κηρύξουν άκυρο το αποτέλεσμα αλλά με κάπως αυθαίρετα πρότυπα για το τι αποτελεί η κατάχρηση, όπως η καταστροφή μιας κάλπης ή η διατάραξη της εκλογικής διαδικασίας μπορεί το 5% των καλπών να καταστραφούν. Και αυτό τελικά να αντιστρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών, εφόσον κάποιοι αποφασίσουν ότι υπήρξε κατάχρηση από πυρανοθείας. Οι κεντρικές εφορευτικές επιτροπές δεν θα μπορούν να ε, ανακοινώσουν τα επίσημα αποτελέσματα λόγω αυτού του νόμου και αυτή τη διάταξη. Επίση υπάρχει ασάφεια στον εκλογικό νόμο για την δυνατότητα να αμφισβητηθούν τα εκλογικά αποτέλεσματα. Αυτό το ανέφερε και η Δόκτωρ Βόλτσου. Είναι ένα πρόβλημα διαρκέ στην Ουκρανία με τα εκλογικά αποτελέσματα εδώ και χρόνια. Είναι περίπλοκε οι διαδικασίε για την προσφυγή, για την αμφισβήτηση δηλαδή του εκλογικού αποτελέσματο. και πολύ συχνά προκύπτουν και διαφορέ μετά τι εκλογέ και στι οποίε ω τώρα δεν έχει δοθεί και λύση τι θα γίνει τώρα στο μέλλον. Οι διεθνείς παρατηρητές των εκλογών θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπόψη τους τα ζητήματα που ανέφερα και ίσως και άλλα τα οποία αυτή τη στιγμή προκύπτουν ε, στην πράξη, στην ίδια τη χώρα. Δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό βάσει των όσων έχουν γίνει ως τώρα οι διεθνείς παρατηρητές να μην ε, μπορέσουν να παρατηρήσουν τις ε, εκλογές της Ουκρανίας Ούτε φαντάζομαι θα τις κηρύξουν ανελεύθερες, παράνομες και αντιδημοκρατικές. Οι διεθνείς παρατηρητές νομίζω ότι θα πούν ότι είναι αξιόπιστες, ελεύθερες και νόμιμες οι εκλογές. Δεν ξέρουμε βέβαια ποιο θα είναι το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά μοιάζει βάσει και των προηγούμενων εκλογικών αποτελεσμάτων στην Ουκρανία ότι τα αποτελέσματα θα είναι κάπου στη μέση της πλάστικας, της ζυγαριάς μάλλον, συγγνώμη. Και η μετακίνηση των ανεξάρτητων βουλευτών θα καθορίσει τελικά το που θα ε, καταλήξει το αποτέλεσμα. Οι παρατηρητές βεβαίως ε, θα μπορέσουν μόνο μέσω της καταμέτρησης του εκλογικού αποτελέσματος να καταλήξουν σε σαφή πορίσματα. Επίσης, ο τρόπος που θα επιληθούν με τα εκλογικέ διαφορέ είναι κάτι που θα καθορίσει την αποτίμησή τους. Στις 28 Οκτωβρίου, λοιπόν, έχουμε τις εκλογές. Θα πρέπει να καταλάβουμε πλήρως πώς διαμορφώνεται το κλίμα τώρα, αλλά να περιμένουμε να ολοκληρωθεί και διαδικασία για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Όλοι συμφωνούν, όπω είπε η Δόκτωρ Βούλτσεκ, ότι οι εκλογέ του 2012 θα είναι ένα πολύ σημαντικό δείκτη τη πολιτική πρόοδου τη Ουκρανία. Επίση, ένα δείκτη για το τι επιφυλάσσει το μέλλον για τι προεδρικέ εκλογέ τη χώρα που πλησιάζουν. Σε γενικέ γραμμέ, ανά τον κόσμο, είναι σύνηθε η εκλογική διαδικασία να παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα Μπορεί μια εκλογική διαδικασία που έχει πάει πολύ καλά, που ήταν εύρυθμη, να ακολουθηθεί από μια που δεν, τα πήγε καλά, που δεν πήγε καλά και το αντίστροφο. Στην Ουκρανία φαίνεται εδώ να υπάρχουν πάντως σοβαρές παναχωρήσεις που προκαλούν ανησυχία και ε, έχουν κρόστο το κόδωνα του κινδύνου για τη διεθνή κοινότητα. Γι' αυτό θα χρησιμοποιηθούν εκλογέ ω δείκτης για το τι πρόοδο έχει επιτελέσει η χώρα αυτή από δημοκρατική άποψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εισβάθος ερμηνεία αυτής της ε, προεκλογικής ε, διαδικασίας. Ε, είμαι βέβαιη ότι αυτό θα αποτελέσει προετοιμασία για τις εκλογές και προετοιμασία για την ερμηνεία των όσων θα συμβούν στις εκλογές. Οι παρατηρήσεις σας λοιπόν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσε Ε, δεν θα αντλήσουμε συμπεράσματα σήμερα. Θα ακούσουμε όμως με ιδιαίτερη προσοχή ό,τι ε, ακουστεί από τους συναδέλφους σήμερα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλερ, διότι ήταν μαζί μου στην Ουκρανία πριν από κάποιες μέρες και θα συνεχίσει και η συνεργασία μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν έχω μία ανακοίνωση διότι σε μία έγκυρη γερμανική εφημερίδα λέγει ότι έχει την έκθεση Κόξ ε, και ζήτησα από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να μου δοθεί και εμένα διότι είναι πάντοτε ατυχές οι βουλευτές να είναι οι τελευταίοι οι οποίοι λαμβάνουν τα σημαντικά έγγραφα οπότε στα πλαίσια αυτά θα ήθελα πολύ να το σημειώσετε και εσείς. Τώρα θα συνεχίσω αγγλικά. Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε παρανόηση, κυριολεκτικά παρανόηση, να πω ευθύς εξ αρχής ότι μετά την επίσκεψή μου με τον συνάδελφο Κόβαλ στην Ουκρανία και εφόσον είχαμε και συνομιλίες με αρκετούς Ουκρανούς αλλά και βάσει των ενδιάμεσων ε, εκθέσεων που έλαβα, πρέπει να πω ότι η κατάσταση της χώρας με ανησυχεί. Με ανησυχεί και μάλιστα σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Νομίζω το θέμα δεν είναι αν θα είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα ή λίγο χειρότερα. Δεν θα είναι ελαφρά και μικρή η διαφορά μεταξύ των δύο εκλογικών διαδικασιών. Εδώ φοβάμαι ότι μπορεί να έχουμε περισσότερα έκτροπα σε σχέση με τις εκλογές του 2010. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με τα μέσα μουσικής ενημέρωσης. Ε, υπήρξε μια αναφορά εδώ, ιδίως την πρώτη ενδιάμεση έκθεση των παρατηρητών της Όντου εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τι πληροφορίε οι πολίτε τι αντλούν κυρίω από την τηλεόραση. Τα μέσα μαζική ενημέρωση και το πόρισμα ήταν σαφέ. Το περιβάλλον ε, ενημέρωση των ε, εκλογών αυτών χαρακτηρίζεται από έλλειψη πολιτική πολυφωνία στην τηλεόραση η ανεξαρτησία πραγματικά ε, απουσιάζει από τους τηλεοπτικούς σταθμούς σε εθνικό επίπεδο και η αγορά δεν είναι ε, αρκετά ανεπτυγμένη. Η πολιτικοποίηση και κατοικοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι εμφανής με τους ε, Παρουσιαστέ να υποστηρίζουν ανοιχτά το καθεστώ. Είναι σοβαρής, σοβαροί περιορισμοί που επιβάλλονται σε προσπαθούν να υψώσουν τη φωνή τους ε, με διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι το πόρισμα τη πρώτη ενδιάμεση έκθεση. Και αυτό αφορά όχι μόνο την TVI, ε, αυτό το σταθμό, αλλά και άλλες, άλλα κανάλια. Αυτό διαφέρει από το τι συνέβαινε την προηγούμενη φορά το 2010. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όλοι μας ήμασταν ευχαριστημένοι με το ευρύ φάσμα έκφρασης ε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, στην Ουκρανία. Αυτό ήδη έχει αλλάξει. Ε, υπάρχει υποβάθμιση και υπάρχει και ο σχετικός νόμος ο οποίο στο νομοσχέδιο που αποσύρθηκε μετά την πρώτη ανάγνωση, όμω είμαι σχεδόν βέβαιο ότι σε περίπτωση που κερδίσουν πάλι την πλειοψηφία η Γιούνταρ ε, στο επόμενο, στην επόμενη Βουλή, θα φροντίσουν να περάσει το νομοσχέδιο αυτό ω μέρο τη προετοιμασία για τι προεδρικέ εκλογέ που είναι πολύ σοβαρέ για τον ίδιο τον Πρόεδρο. Εκείνος αυτό έχει στο νου του και εκεί στοχεύει. Προετοιμάζεται για την επόμενη φορά λοιπόν. Νομίζω το ένα στοιχείο λοιπόν είναι τα μέσα μαζική ενημέρωση. Υπάρχουν τώρα ελλείψει και χάσματα στον νόμο που πολλέ από αυτές και πολλά από αυτά ε, σχολιάστηκαν, αλλά κάποιο από την Εφορευτική Επιτροπή με τον οποίο μιλήσαμε είπε ότι τον νόμο τον έχουν φτιάξει πολιτικοί για τους πολιτικούς. Αυτό ήταν μια πολύ γλαφερή περιγραφή του τι συμβαίνει και κατά την εφαρμογή του νόμου βλέπουμε να υπάρχουν χάσματα και έλλειψεις, ασυνέπειες, σε σχέση με τις κατευθυντηρίες γραμμές λόγου χάρη που απουσιάζουν για τις ε, αρχές τι θεωρείται ε, παραβίαση των κανόνων. Α είμαστε σαφεί. Οι κανόνε του ποινικού κώδικα και του εκλογικού, του νόμου δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι αρμόδιες αρχές δεν θα μπορούν να αναλάβουν δράση λόγω των ε, ασαφιών. Ε, κάτι άλλο που είναι σκανδαλώδες είναι η σύσταση η σύνθεση των εφορευτικών επιτροπών. Και εδώ θα ήθελα να παραθέσω το τι είπε ο πρόεδρο τη Κοινοβουλευτική ε, Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη και τη Αποστολή Παρατήρηση, ο Ελβετό Σοσιαλδημοκράτη Ανδρέα Γκρό. Είπε ότι για τη διαδικασία δημιουργίας εφορευτικών επιτροπών βάσει των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχει επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Είναι μονομερή και μεροληπτική η σύνθεση των ε, εφορευτικών επιτροπών από το τοπικό έω το κεντρικό. Συνήθω αυτό που γίνεται είναι να επιλέγονται διαιτητέ, όχι παίκτε. Και στην ε, ε, Ουκρανία υπάρχουν περισσότεροι παίκτε παρά διαιτητέ κριτέ στι εφορευτικέ επιτροπέ. Αυτό πιστεύω ότι θα αποτελέσει πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα των εφορευτικών επιτροπών. Για την εξαγορά ψήφων, το ανέφερα ήδη, για τον ορισμό βλέπουμε ότι αποφάσεις μπορούν να λάβουν οι αρμόδιες αρχές, ακόμη και για πανομοιότυπες υποθέσεις ε, που πρέπει να κρυθούν, ε, μπορεί να καταλήξουν σε τελείως διαφορετικές, ακόμη και αντικρουόμενες αποφάσεις. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν κάποια καθοδήγηση για το πώς να ερμηνεύονται όλες αυτές οι διατάξεις επίσης δεν υπάρχουν ε, ίσοι κανόνες ε, του παιχνιδιού. Οι κρατικοί πόροι χρησιμοποιούνται υπέρ του κυβερνώντο κόμματο, Αυτό είναι μια πρακτική πολύ διαδεδομένη και σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο εκδηλώσεων που οργανώνται σε πόλεις. Οι εκδηλώσεις ε, ουσιαστικά μετατρέπονται σε κομματικέ υπέρ του κυβερνώντο κόμματο και του υποψήφιου του. Αυτό συνέβη και στις προηγούμενες εκλογές βέβαια, αλλά ήταν κάπω εξισορροπημένη η πρακτική αυτή, γιατί διαφορετικά κόμματα υπερίσχυαν στι διάφορες γωνιές της χώρα. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι αρκετά μονομερή. Και υπάρχουν και κόμματα τα οποία σκοπεύουν να ε, εξαιρεθήσουν τους ε, ψηφοφόρους ώστε να ψηφίσουν και πάλι το κυβερνών κόμμα. Αυτό είναι κάτι το οργανωμένο. Επίσης, από τότε που το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε, η μισή από τους εκλεγμένους αντικαταστάθηκαν. Δεν εξυπηρετούν λοιπόν το στόχο τους, ούτε κάνει φορευτικές επιτροπές. Τα εικονικά αυτά κόμματα έχουν βεβαίως ε, την επίδρασή τους και στις μονεδρικές περιφέρειες, όπου η ψήφος δεν πηγαίνει σε ένα από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα ή σε ένα από τα τρία μεγαλύτερα κόμματα, η ψήφος πηγαίνει σε... στο μεγαλύτερο κόμμα και αυτό ευνοεί συνήθως. Ξέρουμε ποιο είναι αυτό. Τελευταίο σημείο. Δεν υπολογίζω στις δημοσκοπήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή, διότι στην Ουκρανία πρέπει να σκεφτεί κανείς ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας που κάνει τις δημοσκοπήσεις. Ποιος υποκρύπτεται. Και προφανώς εδώ ο στόχο δεν είναι να προωθηθεί απλώ το κυβερνών κόμμα, αλλά να προωθηθούν διαφορετικοί από αυτού που μπορεί πραγματικά να τα πάνε καλά, ώστε να δημιουργηθεί αναταραχή και ε, άγχο και στην ε, αντιπολίτευση. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει την ημέρα των εκλογών. Και από τελευταία παρατήρηση, βεβαίω εφόσον η αντιπολίτευση είναι φυλακισμένη, η επικεφαλής της είναι ε, φυλακισμένη, αυτό είναι κάτι το πρωτάκουστο. Βεβαίως θα υπάρξει ε, αντίκτυπος. Ε, το 2004 ο Γιανοκόβιτς είχε νοθεύσει τις εκλογές αλλά αναγκάστηκε εκ των υστέρων να διευρύνει το πολιτικό φάσμα και να συζητήσει ανοιχτά κάποια πράγματα. Αυτό σήμερα δεν συμβαίνει και βεβαίως ο αντίκτυπο θα είναι τους. Αυτό είναι ήδη ένα δείγμα μέτρηση τη ποιότητα που θα έχουν ε, αυτέ οι εκλογέ στην εξαγωγή του. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερα άτομα έχουν ζητήσει το λόγο και θεωρώ ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλους. Ένας πέμπτος το πολύ. Ο κύριος Σάριος Βόλσκι θα είναι ο τελευταίος και θα κλείσει τη συζήτηση. Έξι τελικά είναι και ο κύριος Ρούτσεκ. Δεν δέχομαι άλλους. Ένα λεπτό, ενάμιση λεπτό ο καθένας για να δώσουμε και πέρα, ε, στη συνέχεια και τη δυνατότητα στις καθηγήτριες να απαντήσει το λόγο. Και κυρία Χάρμς, ε, είμαστε 7 τώρα. Κλείνει ο κατάλογος. Διότι δάλλως δεν θα σεβαστούμε την ώρα και 12 και μισή πρέπει να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση. Θα μπορέσουμε όμως να ξανασυζητήσουμε την Ουκρανία ενώπιση των εκλογών. Ο κύριος Ντάβιτ καταρχάς. Ευχαριστώ. Ετοιμαζόμουν να ψηφίσω αντί να ανοίξω το μικρόφωνο. Δεν θα ψηφίσω για τις ουκρινικές εκλογές, όχι ακόμα. Λοιπόν, καταρχάς να ευχαριστήσω τις δύο προσκεκλημένες μας και τους συναδέλφους ε, για τις εισαγωγικές τους παρατηρήσεις. Ε, θα ήθελα να προσθέσω ένα ε, θέμα ακόμα το οποίο μάλλον δεν αναφέρθηκε. Αναφερθήκαμε σε διάφορες μορφές χειραγώγησης, αλλά δεν αναφέρθηκε η χειραγώγηση από το δικαστήριο και δυστυχώς θεωρώ ότι όλο το δικαστικό σύστημα εργάζεται υπέρ ε, μιας πολιτικής δύναμης. Δεν ε, ξέρω ε, καμία ένσταση η οποία να υποβλήθηκε από κάποιο άλλο κόμμα που να έχει να αποδεχτεί είτε σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο είτε σε εφετείο και θεωρώ ότι αυτό είναι εις βάρος της δημόσιας εικόνας της χώρας και νομίζω ότι αντανακλά το γεγονός ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα κράτος δικαίου τουλάχιστον ε, όχι βάσει των παραμέτρων και των αξιών που θα θέλαμε ε, να συμμερίζεται η Ουκρανία με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε και ο Μάϊκόλ, όταν ε, αναφέρθηκε σε κόμματα πλαστά σε συγκεκριμένες περιφέρειες, είναι αυτό που στην Ουκρανία αποκαλούνται τεχνικοί υποψήφοι. αγοράζονται αυτοί οι υποψήφοι και έχουμε αποδείξεις εδώ στο Κοινοβούλιο για τέτοιες περιπτώσεις και για άλλη μια φορά δυστυχώς τα δικαστήρια δεν έκαναν τίποτα και αυτό είναι λυπηρό. Ε, δεν έχουμε βέβαια αποφασίσει αν θα θεωρηθούν ακόμα δίκαιε ή όχι εκλογέ, ε, δεν γίνεται αυτό εκ των προτέρων, αλλά σε μία από τι διαφάνειε που μα δείξατε, κυρία ε, Βόλτσικ, ε, υπήρχε μία διαφάνεια που αναφερόταν στην ε, ημέρα των εκλογών. Δυστυχώς η διαδικασία είναι μία δημοκρατική διαδικασία και οι διαμαρτυρίε μα είναι για όλη την προεκλογική διαδικασία και είναι λυπηρό ο τρόπο με τον οποίο διεξάγεται. Uh, ο κύριος Τάνοκ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ στην αίθουσα εσείς, εγώ και ο κύριος Άριος Βόλσκι ήμασταν εδώ και το 2004. Και έχω χάσει το λογαριασμό των εκλογικών αναμετρήσεων που παρακολούθησα ε, στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτός, αυτές οι συγκεκριμένε θα είναι αποφασιστική σημασία για τη γεωπολιτική σημασία αυτής της πολύ μεγάλης χώρες. Θα πάει προς την... Ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα πάει προς την ε, ρωσική πλευρά και θα ζητήσει στήριξη από αυτούς. Από στρατηγική πλευρά, λοιπόν, εξετάζουμε κατά πόσον θα είναι ελεύθερε και δίκαιε αυτέ οι εκλογέ ε, βάσει των διεθνών κανόνων. Και θα ήθελα να ρωτήσω την ε, καθηγήτρια Μπέρτ, καταρχά. Υπάρχει κάποιο προηγούμενο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ε, για να ε, δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στις ε, αποστολές παρατήρησης εκλογών για να εξετάσουμε κάποιες εκδοχές για το κατά πόσον έχουν γίνει επιλεγμένες κατηγορίες για προσφυγή στα δικαστήρια κατά υποψηφίων της αντιπολίτευσης. Έχουν διαπιστωθεί κάποια περιστατικά από διεθνείς παρατηρητές σε άλλες περιοχές, διότι ποτέ στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια δεν ξέρω κάτι ανάλογο. Προς τον αγαπητό συνάδελφο από την ομάδα μου τώρα, κύριε Ντάβιτ, ε, παραδοσιακά στις χώρες του ΑΣΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον είναι ίσον σημασία. Ε, το 2004, στον ε, τριαδικό σχηματισμό που είχαμε την ε, ε, κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη συμμετοχή του ΑΣΑ, το ΑΣΕ. Ε, εκεί συνήθω ο ΑΣΕ είναι αυτός ο οποίος έχει τον κύριο ρόλο και εμείς είμαστε στα μετόπισθεν. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι ε, κακό όπως ήταν και το 2004 που κάποιοι προσπαθούσαν να πιέσουν τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογιών ε, ε, βγήκε νικητής ο Γιαννουκόβιτς ενώ ήταν σαφές ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν ο νικητής. Ε. Εσείς ε, διατηρείτε το δικαίωμα ε, να ετοιμάσετε ξεχωριστή έκθεση αν θεωρήσετε ότι η εκλογική διαδικασία δεν προχώρησε όπως έπρεπε να γίνει. Υπάρχει κάτι τέτοιο Το Έχω θίξει και στα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ε, και το θίγω και εδώ σήμερα. Θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα από πολιτική σκοπιά και το επιτρέπουν και οι κανόνε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν χρειαστεί να υπάρχει ξεχωριστή έκθεση από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι εκλογέ. Ah. One minutes, I think we have. 1,5 λεπτό νομίζω σας είπαμε, αλλιώς ε, θα καθυστερήσουμε διότι είναι ήδη 12 και τέταρτο. Ο κύριος Σεβερίν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που διοργανώσετε τη συγκεκριμένη ακρόαση, είναι πολύ χρήσιμη. Πολλές πληροφορίες και θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε βεβαίως αυτές τις πληροφορίες, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε ε, οπωσδήποτε να δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι έχουμε εξαγάγει τα συμπεράσματά μας πριν ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία. Συμφωνώ μεν ότι οι εκλογές είναι μια όλη διαδικασία και δεν είναι μόνο μια ημέρα, αλλά τα συμπεράσματα εξάγονται στο τέλος της διαδικασίας. Και αυτό είναι σημαντικό για να προσδώσει και αξιοπιστία στα συμπεράσματά μας. Δεύτερον, θεωρώ ότι ε, είναι λογικό να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας και τις αμφιβολίες μας ως έγκαιρη προειδοποίηση. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που μας ανησυχούν και θα πρέπει δικαίως να ζητήσουμε από τις αρμόδιες αρχές να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να βελτιώσουν την κατάσταση όσο μπορεί να βελτιωθεί για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Επιπλέον, θα ήθελα να προσθέσω και το γεγονός ότι στο τέλος θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι, να κάνουμε μια αμερόληπτη αξιολόγηση, αλλά δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι είμαστε πολιτικοί και ότι έχουμε και γεωπολιτικά συμφέροντα και τα συμπεράσματά μας, τα οποία πρέπει να είναι δίκαια, θα πρέπει να είναι συνεπή και προς τις ε, γεωπολιτικές ε, και πολιτικές μας ε, επιλογές και το θεματολόγιό μας. Και τέλος, μια τελευταία παρατήρηση, επιτρέψτε μου, ναι, μεν πολλά προβλήματα, πάρα πολλές αδυναμίες, αλλά δυστυχώς κάποιες από αυτές τις δυναμίες θα μπορούσαν ίσως σε μικρότερο μέγεθος, σε ε, μικρότερες τάξεις μεγέθους να αναγνωριστούν και στις χώρες μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να τα βλέπουμε όλα με ένα ε, πρίσμα πιο ε, σχετικό. Ευχαριστώ. Εφόσον έχω 1,5 λεπτό, έχω μόνο ερωτήσεις. Προς την δόκτωρα Βόλτσουκ κυρίως. Αναφέρατε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Τι ρόλο θα έχουν μετά τι εκλογέ. Πρώτον. Δεύτερον. Αναφέρατε το τι συμβαίνει με την αντιπολίτευση. το Γιούνταρ ανεβαίνει, ιδίω ο επικεφαλή. Πώς το εξηγείτε. Τι γίνεται όμως εάν ε, σκεφτούμε ότι η Τιμοσέγκο είναι στη φυλακή στην Ουκρανία φαίνεται ότι υπάρχει μια κόπωση από αυτή την τόσο επιθετική συμπεριφορά και ε, την τόσο αρνητική τοποθέτηση της ε, Fatherland, του Fatherland. Μ' άρεσε πάρα πολύ επίση ε, ο χάρτη σα με τι εθνικέ μειονότητε. Αλλά πώ εξηγείτε την κατάσταση, Είναι 12.000 οι Ρώσοι φυσικοί ομιλητέ σε μια χώρα 36 εκατομμυρίων. Υπάρχουν βεβαίω και ομιλητέ ε, τη Ουκρανική. Υπάρχει το κόμμα των περιφερειών στο Νότο, όμω η πλειοψηφία στι τελευταίε εκλογέ, δείτε και τι δημοσκοπήσει και την αποτύπωση τη κατάσταση στι μονεδρικέ, φαίνεται ότι το ίδιο θα συμβεί και πάλι. Το κόμμα των περιφερειών πάλι θα νικήσει. Γιατί πιστεύετε ότι το ψηφίζουν οι άνθρωποι τελικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά τη γνώμη μου ένα είναι σαφές σχετικά με την ε, παρατήρηση αυτών των εκλογών θα πάμε με μία, ένα μακρύ κατάλογο από αμφισβητήσεις και προβλήματα που δεν χρειάζεται να συγκαλύψουμε. Δεν μπορεί ε, να καταλήξουν οι εκλογές αυτές όπως ε, αξιολογήθηκαν σε προηγούμενα χρόνια οι εκλογές στην Ουκρανία και, η Ουκρανία και πρέπει να είμαστε σαφείς. Όσον αφορά τον Πατκόφς και τον η το θέμα δεν έχει καμία σχέση με τις εκλογές ε, ήταν ε, ανθρωπιστική αποστολή για να αξιολογήσουν ε, την κατάσταση των φυλακών αλλά κατέληξε κατευθείαν σε συμπεράσματα που είναι σημαντικά πέραν από την εντολή με την οποία μετέβησαν δηλαδή και για τα θέματα των εκλογών και θα επηρεάσουν την αξιολόγηση των συνθήκων διεξαγωγής των εκλογών. Φοβούμε λοιπόν ότι σε συνεργασία με τα αποτελέσματα του ταξιδιού του κυρίου Γκάλερ και του κυρίου Γκάλερ μπορεί αυτά να παραποιηθούν και ενδεχομένως η κατάσταση ε, στην, ε, ε, στην Ουκρανία θα πρέπει να διευκρινιστεί. Επιπλέον πρέπει να δούμε ε, εάν ε, υπάρχει μία γεωπολιτική ε, σχέση δηλαδή για να δούμε προς ποια κατεύθυνση κατευθύνονται οι Ουκρανοί θα στραφούν προς τη Ρωσία ή προς τη Δύση εγώ αξιολογώ ότι η χώρα αυτή πρέπει να έχει καλές σχέσεις, λειτουργικές σχέσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις βασικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αυτό δεν σημαίνει σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει κάνει μία πρόταση με την ε, Συμφωνία Συνεργασίας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως σας είπα δεν θα δεχθεί, και ε, θα δεχτεί ε, καταστάσεις οι οποίες δεν είναι δημοκρατικές. Ο κύριος Ζάιρος Βόλσκι. Τρει ερωτήσει έχω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτον, γιατί, νομίζω η κυρία Μπέρτς το είπε, ηγέτες στη φυλακή θα είναι νόμιμες εκλογές. Ερωτηματικό βάλατε. Γιατί βάζετε ερωτηματικό, ρωτάω εγώ. Εάν είναι επιλεκτική δικαιοσύνη και βάζαμε τον Ομπάμα ή τον, ε, τον άλλο στη φυλακή, θα θεωρούσατε τις αμερικανικές εκλογές και την αμερικανική δημοκρατία ε, ε, ευρύθμος λειτουργόσα. Επίσης η απόφαση η έκθεση Κόξ ε, Κρασνιεύσκη να αποκριθεί, να αποκριθεί είναι λανθασμένη. Και τρίτη ερώτηση για τις μονεδρικές. Ένα από τα αποτελέσματα που ακούσαμε, από τα συμπεράσματα που ακούσαμε είναι ότι η αντιπολίτευση ήταν πιο αδύναμη στις μονεδρικές από ό,τι στις αναλογικές. Αυτό γιατί βασιζόμαστε στο ότι το κόμμα, το υποψήφι Γιούνταρ και Φάδερλαντ δεν θα είναι κοινοί υποψήφοι, θα, κατέβουν ξεχωριστά. Αν όμως συμφωνήσουν σε κοινούς υποψηφίους, πώς θα επηρεαστούν τα αποτελέσματα. What implication... Και τρίτη ερώτηση. Τι επιπτώσεις θα έχουν αυτές οι άδικες εκλογές, τις προεδρικές, το 2015. Το παιχνίδι έχει ήδη αρχίσει. Ευχαριστώ. πολύ. Και τώρα οι δύο μιλήτριες. Αντίστροφα θα λάβουν το λόγο. I'm uh, thank you very much. I'll take... Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις παρεμπιπτόντως. Πολύ ενδιαφέρουσες. Για την ερώτηση για τους ηγέτες. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αν αυτές ήταν προεδρικές εκλογές και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης ήταν στο φυλακή, θα ήταν τελείως διαφορετικό το ζήτημα. Αλλά επειδή οι εκλογές αυτές είναι κοινοβουλευτικές και το κόμμα της κυρίας Τιμοσέγκο ούτως ή άλλως αμφισβητεί τις εκλογές, όπως σας είπα και προηγουμένως, το ερώτημα είναι ως ποιο βαθμό η δυνατότητα ενό κόμματος να αμφισβητεί ε, τις εκλογές ε, σχετίζεται με το γεγονός ότι αυτή και αρκετά μέλη του κόμματός τη είναι στη φυλακή και η ίδια δεν είναι σε ε, θέση να αμφισβητήσει ε, την, τις εκλογές για το Κοινοβούλιο. Όπως σας είπα, είναι σοβαρό πρόβλημα. Πέρα από τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεων που μπορούν να εξεταστούν και μεμονωμένα, δεν αφορούν μόνο τις εκλογές. Ε, το όλο θέμα της διεξαγωγής της ε, εκλογές, ε, εγώ θεωρώ ότι εδώ όντως διακυβεύεται. Επειδή όμως δεν είναι προεδρικές οι εκλογές, δεν δίνεται ουσιαστικά δικαίωμα να απαρατήτως να πούμε ότι μπορούμε να αμφισβητήσουμε όλη την εκλογική διαδικασία. Εγώ δεν ξέρω κάποιο συγκεκριμένο προηγούμενο, με ρωτήσατε, το σκεφτόμουν μάλιστα και πριν έρθω εδώ. Έχει υπάρξει προηγούμενο πολιτικών που έχουν ε, φυλακιστεί και δεν είναι σε θέση να αμφισβητήσουν τις εκλογές, αλλά ε, υπάρχουν τρεις πτυχές σε αυτή την περίπτωση. Καταρχάς είναι ο νόμος, που νομίζω ότι αυτό, είναι, αυτό που μας ανησυχεί λιγότερο. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και δεν έχουν κάτι τέτοιο ε, στη νομοθεσία τους. Παραδείγματος χάρη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν κάποιος είναι φυλακισμένος δεν έχει εκλογικά δικαιώματα. Δεν λέω λοιπόν ότι είναι θέμα νόμου, δεν λέω ότι είναι αποδεκτή βέβαια η πρακτική, αλλά ε, ο νόμος δεν είναι αυτό που μας ανησυχεί τόσο πολύ. Η βασική ανησυχία είναι γιατί εγκρίθηκε μια τέτοια νομοθεσία και ε, από εκεί και πέρα για τις διάφορες μεμονωμένες περιπτώσεις ε, ε, και το γεγονός ότι η δικαιοσύνη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μάλλον επιλεκτική. Αυτά είναι πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβή παραλληλισμό μεταξύ χωρών, διότι σε κάθε χώρα ε, τα πάντα εξαρτώνται από τις συνθήκες. Στην Ουκρανία μπορεί να υπάρχει, ε, να γίνει μια σύγκριση και να δούμε ότι είναι αντίστοιχη νομοθεσία σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε μια άμεση σύγκριση με το τι κάνουν άλλες χώρες και τι νομοθεσία έχουμε. Θα πρέπει να δούμε την όλη πορεία της ε, διαδικασίας στην Ουκρανία και νομίζω ότι αυτό είναι το μοναδικό στην περίπτωση της Ουκρανίας. Τώρα, για τι ε, μονοιδρικέ περιοχές και για το κατά πόσον το ΟΥΝΤΑΡ και το Φάδερλαντ θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και κατά πόσον αυτό θα αποτελέσει μειονέκτημα, νομίζω ότι οι περισσότεροι ε, σχολιαστές και παρατηρητές Κατά πάσα πιθανότητα, βασισμένοι και στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, θα πούνε ότι υπήρχε μειονέκτημα διότι υπήρχε το όλο θέμα της ε, κατάχρησης των διοικητικών πόρων από το κυβερνών κόμμα. Ε, τους έδινε ένα πλεονέκτημα ιδίω στις μονοεδρικές περιφέρειες και γι' αυτό ε, πολλοί ανησύχησαν με την ε, επανένταξη αυτών των μονοεδρικών περιφερειών στην ε, Ουκρανία. Και τους ανησύχησαν φυσικά και ανησύχησαν ιδιαίτερα και τις εκλογές του 2002. Γι' αυτό λοιπόν ανησυχεί πολύ η κατάσταση. Όχι τόσο το τι θα προτιμήσει ο κόσμος και τι θα επιλέξει, αλλά το, τις πρακτικές που χρησιμοποιεί το κυβερνών κόμμα, χρησιμοποιεί διοικητικούς σπόρους για να επηρεάσει την προτιμήσή τους. Νομίζω λοιπόν ότι συντρέχει λόγος ανησυχίας ε, πέραν από την ικανότητα της ε, αντιπολίτευσης να συνεργαστεί. Από εκεί και πέρα η κυρία Βόρτσικ θα σας πει ε, τι, συνέ, τι συνέπειες υπάρχουν για τις εκλογές του 2015. Παρακαλώ. Πραγματικά συναρπαστικέ οι παρατηρήσεις σα, ε, πολύ ευστοχέ, αλλά θα αναγκαστώ να είμαι πολύ επιλεκτική και ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη. Για το θέμα τη πολυφωνία στα μέσα μαζική ενημέρωση. είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ τη διαρθρωτική δομή, τη. Ε, Ουκρανίας και το τι συμβαίνει με τις καταχρήσει και τις παραβιάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωση. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα μέσα μαζικής ενημέρωση. Κάποια τηλεοπτική σταθμή είναι κρατική ιδιοκτησία. Η δομή του είναι πολύ σαφή και η Ουκρανία δεν έχει κανάλια δημόσια. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχουν ίσοι κανόνε παιχνιδιού για όλε τι πολιτικέ δυνάμει. Αυτό όμω πολλαπλασιάζει τον αντίκτυπο των προβλημάτων. Υπάρχει η λογοκρισία και από την άλλη οι διαρθρωτικέ ε, ιδιαιτερότητε που ουσιαστικά εντείνουν τι πολιτικέ δυσκολίε. Επίσης το θέμα της χαμηλής ποιότητας των ίδιων των νόμων συμπεριλαμβανομένου του εκλογικού. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο στην Ουκρανία. Είναι συχνό. Οι νόμοι γράφονται από τους πολιτικούς για να ψηφιστούν και να ωφελήσουν τους πολιτικούς με πολλές ασυνέπειες και πολλά παραθυράκια. Όμως αυτό που είναι σημαντικό για την Ουκρανία και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το, να κρατήσουμε στο μυαλό μας πριν τις εκλογές, είναι πώς καλύπτονται αυτά τα παραθυράκια, πώς χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν πολλέ τεχνικέ δυσκολίε. Υπάρχει όμω τρόπο να επιληθεί το ζήτημα με τα παραθυράκια με τρόπο δίκαιο και νόμιμο ή ωφελείται ένα, το ένα από εις βάρος του άλλου κόμματο. Είναι ένα σημαντικό δείκτη αυτό για την ποιότητα των, εκλογικών αυτών, των εκλογών αυτών καθεαυτών. Επίση, το πολιτικό κλίμα, οι εντάσει, η δυσφορία τη αντιπολίτευση είναι σημαντικά. Φαίνεται να... Σημαντικά στοιχεία. Φαίνεται να επιβάλλονται κυρώσει κατά τη αντιπολίτευση ή να επιτρέπεται η συμμετοχή στι εκλογέ με τρόπο πολύ συγκεκριμένο. Η πολιτική δράση πάντοτε δημιουργούσε προβλήματα στην Ουκρανία και πάντοτε οι κυβερνώντε προσπαθούσαν να προβλέψουν τι κινήσει των αντιπάλων του. Πάντοτε υπήρχαν τεχνικέ ε, δυσκολίε, πάντοτε υπήρχαν διαφωνίε. Πώ επιλύονται. Μια άλλη διαθωτική δυσκολία στην Ουκρανία είναι το δικαστικό σύστημα ο δικαστικό κλάδο δεν είναι ανεξάρτητο και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα έχει και αποτέλεσμα στη αντίκτυπο την ποιότητα των εκλογών. Όμω υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαδοτικών ιδιαιτεροτήτων και πώ χρησιμοποιούνται από τι πολιτικέ δυνάμει. Τώρα για το Κομμουνιστικό Κόμμα, πολύ σύντομα. Είναι αξιοσημείωτη η αναβίωσή του. Ε, ουσιαστικά θεωρήθηκε ένα κόμμα των συνταξιούχων κάποια στιγμή αλλά σκοπός είναι να μαζέψει ψήφους από τους αποκοτευμένους ψηφοφόρους στην Ανατολική και Νότια Ουκρανία οι οποίοι θα είχαν ψηφίσει το κόμμα των περιφερειών. Επειδή όμως υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, μάλλον δεν θα συμβεί αυτό το κομμουνιστικό λοιπόν κόμμα. Για τους απογοητευμένους, αγανακτισμένους ε, ψηφοφόρους, σε περιφέρειες όπου ήταν ε, πάντοτε τα οχυρά του κόμματος των περιφερειών, υπάρχουν σοβαρές ελπίδες δεν σημαίνει ότι το κόμμα Φάδρελαντ, η Γιουντάρ, θα θα έχουν ένα σοβαρό συνομιλητή απέναντί του με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα μπορούσε στο παρελθόν να συνεργαστεί και με το Κόμμα των Περιφερειών. Μάλιστα στο παρελθόν είχε καλύτερη σχέση με τα κόμματα της Νότιας και Ανατολικής Ουκρανίας. Αυτή είναι η μόνη πρόβλεψη που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Γιούνταρ τώρα είναι ένα κόμμα που δείχνει την κόπωση που υπάρχει με τις πολιτικές συγκρούσεις γενικώ. Θα μπορούσε να είναι μια φρέσκια δύναμη, μια νέα πνοή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και έχει και μια πολύ καλή εκλογική προεκλογική εκστρατεία. Ε, έχει πολύ ισχυρή επίση ε, αντιπροσώπευση στην πρωτεύουσα. Επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη ε, απογοήτευση στην πόλη του Κιέβου, επειδή είναι άμεση επαφή με την πολιτική ελίτ, γι' αυτό και υπάρχει τέτοια μεγάλη επιτυχία. Δημιουργείται ένα τέτοιο πολιτικό κλίμα με μια ιδιαίτερη πλατφόρμα, διότι η συμμετοχή στο Κοινοβούλιο θα είναι πολύ σημαντική για οποιονδήποτε υποψήφιο των προεδρικών εκλογών. Περιθωριοποιείται πολύ εύκολα οποιοδήποτε υποψήφιο δεν καταφέρει να έχει μια έδρα στο Κοινοβούλιο. Και για τη συμμετοχή του στην προεδρική προεκλογική εκστρατεία, αλλά και για το κατά πόσο μπορεί να αντιστρέψει το αποτέλεσμα του, που είναι συνήθω υπέρ του κυβερνώντο. Κύριε Κόβαλ, ευχαριστώ. Σχόλια για την ερώτηση του κυρίου Τάνοκ για το πώς θα δουλέψουμε, ποια θα είναι η μεθοδολογία μας. Διαρκώς έχουμε επαφές με τους επικεφαλείς της αντιπροσωπείας του ΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το ΝΑΤΟ δεν έχει φτάσει ακόμη στην Ουκρανία, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η στάση τους. Όμως, από μια σύντομη παρατήρηση της κατάστασης, ξέρουμε ότι η συνεργασία θα είναι αρμονική. Για τις νομικές πτυχές, θα ζητήσω μια νομική ανάλυση από τις νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου για να δούμε τι θα μπορούσε να συμβεί τι δυνατότητες υπάρχουν να συντάξουν μια ξεχωριστή έκθεση. Ως προς τα θέματα ουσίας, νομίζω είδαμε ε, διαβίου, δια, ε, Είδαμε τους σύνεγγυς με την, επιτροπή, με την αποστολή του ΟΑΣΕ το τι συμβαίνει στη χώρα και χρησιμοποίησαμε συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα μπορούσε να ξαναχρησιμοποιηθεί. Όμω η εκλογική διαδικασία δεν θα είναι το μόνο στοιχείο το οποίο θα αποτιμήσουμε. Θα είναι η ίδια η προεκλογική περίοδο, η διεξαγωγή των εκλογών, η ανάληψη τη εξουσία. Ίσως να μην βρισκόμαστε βέβαια εκεί, διότι λόγω του πολιτικού συστήματος ε, θα καθυστερήσει αυτό. Αλλά βασικός στόχος είναι να βασιστούμε στη μεθοδολογία του ΑΣΕ, οι οποίοι έχουν πολύ συγκεκριμένε γνώσει, πολύ συγκεκριμένε πρακτικέ και θα τι αξιοποιήσουμε. Το θέμα είναι σε τι βαθμό τα συμπεράσματά μα θα αντικατοπτρίζουν το πολιτικό σκηνικό, όπω είπε ο κ. Εβερίν, και κατά πόσον θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε περισσότερο τεχνικέ παρατηρήσει. Κάθε μια από τις δύο επιλογές θα έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις. Ένα τεχνικότερο περιεχόμενο, εφόσον ασχοληθούμε με τα αποτελέσματα των εκλογών περισσότερο, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει και τις απόψεις διάφορων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, ε, διότι όπως είπε η Άστον, ε, είναι πολλές πολιτικές ομάδες και οι χώρες που θα τοποθετηθούν σχετικά. Η αντιπροσωπεία μας νομίζω ότι θα βρίσκεται σε πολύ καλή πολιτική θέση. Ο αντιπρόεδρος ε, των ε, Πρασίνων θα βρίσκεται μαζί μας, ε, επίσης της ε, Επιτροπής ΑΦΕΤ. Είμαστε όλοι επαρκώς καταρτισμένοι, δεν υπάρχει φόβος και δεν νομίζω ότι υπάρχουν και διαφωνίες για το τι συνεργασία μπορεί να έχουμε μεταξύ μας, αλλά και με τα μέλη της αποστολής του ΑΣΕ. Ο χρόνος θα δείξει. Ο χρόνος θα δείξει τι θα γίνει στο μέλλον. Ελπίζω ότι θα υπάρχουν νομικές εγγύσεις. Κύριε Τάνοκ, να σας ευχαριστήσω για το σχόλιο σας. Πόση ανεξαρτησία θα πρέπει να έχουμε εμείς οι ίδιοι και τι συνέπειες θα υπάρξουν για τις μελλοντικέ αποστολές παρατήρησης. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Θα ζητήσω τις συμβουλές σας και πριν τις συναντήσεις μας στο Κίεβο και το πόρισμά μας θα εξαρτηθεί από την επόμενη των εκλογών ημέρα. Αυτό τότε θα κρυθούν όλα. Δεν θα ήθελα τώρα να κάνω αυστηρά σχόλια επικριτικέ παρατηρήσεις, διότι τα σχόλιά μας μετά τις εκλογές θα είναι νομίζω πιο εύστοχα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κόβαλ, τις ε, πυρογνώμονές μας. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια αξιολόγηση. Θεωρώ ότι μια αποστολή δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται απλώς και μόνο στις τεχνικές πτυχές των εκλογών. Θα πρέπει να επαληθεύσουμε και πώς ε, πήγε η όλη εκλογική διαδικασία, ε, να λάβουμε υπόψη ε, όλο το πλαίσιο. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια συνολική εικόνα. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πάντα υπήρχαν λήψεις, ε, κενά, προβλήματα. Το 2005 υπήρχαν περιστατικά νοθείας ε, στις εκλογές εκεί και αυτοί οι οποίοι ε, είναι υπεύθυνοι δεν κατέληξαν στη φυλακή, αλλά ήταν και πάλι υποψήφοι. Ενώ αυτοί οι οποίοι ήταν υποψήφοι στις προηγούμενες εκλογές ε, είναι τώρα στη φυλακή. Πρόκειται λοιπόν για διαφορετικής φύσεως προβλήματα και θα πρέπει να γίνουν ποιοτικέ διαφοροποίησεις στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε την κατάσταση. Θα πρέπει επίσης να ε, έχουμε κατά νου και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Νοεμβρίου, στις 25 Νοεμβρίου του 2010 υπήρχε αυτό το ψήφισμα, για τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές ε, επί τη βάση των όσων ε, είπαν οι επιροχνόμονες ε, στις εκλογές εκείνες η αντιπολίτευση, η κυρία Τιμοσέγκο και όλοι οι υπόλοιποι δεν μπόρεσαν καν να υποστηρίξουν τους υποψηφίες τους. Και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε σαφέστατα ότι πρόκειται για υπιστοδρόμηση, πολύ σοβαρή οπισθοδρόμηση, σε σχέση με τις ε, κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές του 2006 και του 2010. Δεν θα πρέπει λοιπόν ε, να λησμονούμε και το εν λόγω ψήφισμα. Φυσικά κανείς δεν είναι ε, αναμάρτητος, ε, υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν θα πρέπει να σιωπούμε. Θα υπάρχουν και ποιοτικέ διαφοροποίησεις. Δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε λοιπόν μόνο στις τεχνικές πτυχές της διεξαγωγής των εκλογών, θα πρέπει να σκεφτούμε και τι ελπίδες έχει η αντιπολίτευση. Ένα μεγάλο τμήμα της αντιπολίτευσης ε, είναι στη φυλακή. Ε, μέλη των υποψηφίων στη, τοπικά και περιφερεια... στις τοπικές και περιφερειακές αρχές αντιμετωπίζουν σωματικές δυσκολίες, πιέζονται από διοικητικές υπηρεσίες υπηρεσίε, από δικαστήρια και όσον αφορά την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης εν γέννη, το Υπουργείο Οικονομικών και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός είναι ε, οι ιδιοκτήτες των βασικών τηλεοπτικών σταθμών. Είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι αυτά είναι ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να μην μιλήσω δε για το TV1. Ε, άλλαξαν οι συχνότητες, ε, τώρα πλέον δεν διατίθεται ε, μέσω καλωδιακής τηλεόρασης και δεν μπορεί κανείς να δει το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο. Επομένως, θα πρέπει να γίνει και μία λογική αξιολόγηση. Πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουμε τα πράγματα γενικά. Δεν μπορούμε βέβαια να προδικάσουμε τα αποτελέσματα και να είμαστε προκατηλημένοι για αυτές τις εκλογές, γιατί θα τεθεί και θέμα αξιοπιστίας. Και εάν δεν μπορούμε εμείς να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία μας στις αποστολές παρατήρησης εκλογών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σίγουρα θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Επομένως, η αντιπροσωπεία παρατήρησης των εκλογών. Τη Δευτέρα το πρωί θα συζητήσει όλα αυτά τα ζητήματα. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Κόξ και τον κύριο Κρασνιεύσκη που έχουν και μία έκθεση για τις δικές τους αποστολές. και θα μιλήσουμε και για τα όσα είπε ο ε, Αναφερόμαστε σε επιλεκτική δικαιοσύνη και σε εκλογές ε, στη συγκεκριμένη έκθεση και θα είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τις ε, φιλοξενούμενές μας, ευχαριστώ τους συναδέλφους και καλή σας ημέρα.